δίκαιο κοινωνικά να πούμε πως όταν μια επιχείρηση απασχολεί 5.000 άτομα είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει, για να φαλυρίσει, επεμβαίνει το κράτος, δεν ξέρουμε ποια μορφή, μέχρι στιγμής είναι κρατική συμμετοχή. Αλλά είναι δίκαιο ταυτόχρονα να αφήσουμε 50 επιχειρήσεις με 100 υπαλλήλους κάθε μία να χρεοκοπήσουν και να μην ασχολείται. Μιλάμε για τον ίδιο αριθμό θέσεων τελικά εργασίας είναι ακριβώς πάλι 5.000 άτομα. Γνωρίζω βεβαίως πως υπάρχουν και οι νόμοι της πολιτικής, τους οποίους δεν μπορούμε να, να αγνοήσουμε. Το συμπέρασμα όμως πρέπει να είναι το, το εξής. Δεν είναι ότι πρέπει να σταματήσει να βοηθάει τις μεγάλες επιχειρήσεις ε, η πολιτική, απλά να βοηθήσει τις συνθήκες, το πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να έχουν ευκαιρίες. Αυτή η αρχή του Think Small First. Νομίζω εκεί πέρα ε, βασίζεται και είναι μεγάλη επιτυχία το ότι καταλήξαμε σε αυτή την, την αρχή. Κυρίες και κύριοι, εάν ε, ανακεφαλαιώσουμε το τι κάναμε τα, τα τελευταία χρόνια, ανέφερα το πακέτο της εσωτερικής αγοράς, καταλήγουμε σε έναν πολύ εντυπωσιακό κατάλογο ε, σημαντικών ε, πρωτοβουλειών και αλλαγών για τις οποίες πιστεύω ότι πληρούν και ανταποκρίνονται στις αρχές τις οποίες ανέφερα. Για το πακέτο της εσωτερικής ε, αγοράς θέλω να πω πως κατά την ε, πραγματοποίηση του πακέτου αυτού θα έχουμε και πολύ καλύτερη επιτήρηση της αγοράς στην, εφαρμογή αυτού του πακέτου για να έχουμε και ασφάλεια στην ιστορική αγορά. Και βεβαίως η Επιτροπή, η Επιτροπή σας έχει συζητήσει σε σχέση με το πακέτο της ιστορικής αγοράς το θέμα του σήματος CE. Πράγματι η Κομισιόν έκανε μία μελέτη το συζητήσαμε και με τον συγητή σας και καταλήξαμε από κοινού στο συμπέρασμα πως ε, δεν θα λύσει ένα νέο πανευρωπαϊκό σηματάκι τα προβλήματα τα οποία έχουμε, οπότε καλύτερο είναι να επικεντρωθούμε στο σήμα ΣΕ και να ενισχύσουμε το υπάρχον ε, σύστημα. Επίσης, ε, ασχοληθήκαμε με την ασφάλεια των ε, παιχνιδιών και δημιουργήσαμε μια σύγχρονη οδηγία γιατί είχε φτάσει επιτέλους ε, ο καιρός γιατί τα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα της αγοράς γίνονται λόγω της παγκοσμιοποίησης πολύ μεγαλύτερα. Επίσης ε, δημιουργήσαμε επαναστατική νομοθεσία για τους ε, εξοπλισμούς. Ε, πριν από τέσσερα χρόνια κανείς δεν φανταζόταν κάτι τέτοιο, το καταφέραμε όμως και σε χρόνο ρεκόρ. Και πράγματι ήταν και η πίεση της Επιτροπής σας ε, και της Προέδρου σας που οδήγησε στον εξυγχρονισμό του σχετικού ευρωπαϊκού δικαίου και σκέφτομαι και αυτό το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες ε, με τους πυροπολισμούς σε ένα γερμανικό σχολείο. Σκέφτηκα πόσο ε, καλά τελικά τα καταφέραμε, γιατί θα είχαμε κατηγορηθεί για αμέλεια εάν δεν είχαμε κάνει αυτό που έκαναμε. κάναμε και δεν ξέρω αν επαρκούν και όλες. Γιατί έχω τελικά αμφιβολίες γνωρίζοντας πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερα τα πράγματα με ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί αυτά τα οποία πρέπει να βελτιωθούν είναι κατ' ουσίαν ε, αρμοδιότητα του εθνικού δικαίου και δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Απλοποιήσαμε λοιπόν και το, το το σχετικό δίκαιο. Και επίσης και όσον αφορά τη μετρολογία οδηγηθήκαμε σε κάποιες απλοποιήσεις. Ξέρετε υπάρχει ανεκδοτολογία σχετικά με το, το pint και το mili και τις αγγλικές μονάδες μέτρησης. Αλλά εντάξει αυτά αποτελούν και στοιχεία του πολιτισμού και της ε, ποικιλίε που πρέπει να συμβαστούμε στην Ευρώπη. Να έρθω τώρα στην αυτοκινητοβιομηχανία. να πω το εξή. Και εδώ πέρα νομίζω μπορούμε να θεωρούμε αυτούς ε, τυχερούς για το ότι μαζί με το Cars 21 συζητήσαμε πάρα πολύ νωρίς το ποιο θα είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Και τώρα ε, εν μέσω της ε, κρίσης δεν τίθεται το ερώτημα γιατί το έχουμε ήδη απαντήσει. Το Cars 21 είναι η απάντηση στο ποιο είναι ο δρόμος προς το μέλλον. Η κρίση θα επιταχύνει αυτά τα οποία αναφέρονται στο Cars 21, δηλαδή να γίνει πιο αποδοτική ε, του κόσμου η ευρωπαϊκή αυτοκινητομηχανία, καθώς αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, φιλικότητα προς το περιβάλλον, ασφάλεια και ποιότητα των αυτοκινήτων. Βεβαίως πλήττεται ιδιαίτερα από την κρίση η ευρωπαϊκή α, ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά εντάξει, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει πλήττεται από την ε, κρίση. Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση για το ότι θα επιζήσουν όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από αυτή την κρίση, αλλά εγώ θα το διατύπωνα αλλιώς. Δεν υπάρχει και αναγκαιότητα να πούμε πως πρέπει να εξαφανιστεί κάποιος Ευρωπαίος ε, κατασκευαστής γιατί είναι όλοι οι κατασκευαστές τόσο καλοί που μπορούν να συνεχίσουν να ε, υπάρχουν. Επίσης σε σχέση με την κρίση της General Motors θα πρέπει σύντομα να λάβουμε κάποιες ε, αποφάσεις, όχι ακόμα όμως, γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση μέχρι να ξέρουμε ποιο είναι το συνολικό μέλλον της επιχείρησης και αυτά τα οποία ακούσαμε το Σαββατοκύριακο από την Ουάσιγκτον που έγινε πιο συγκεκριμένα σήμερα μία ανακοίνωση του Πρόεδρου του κ. Ομπάμα για εμένα σημαίνουν ότι οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν την αυτοκίνητομηχανία τους να διαλυθεί. Οπότε για εμάς σημαίνει πως εξακολουθεί να υπάρχει ευθύνη της General Motors για τις ευρωπαϊκές θυγατρικές. Και τους λέω εγώ παντού δεν μπορείτε να απαλλάξετε General Motors από την ευθύνη της για την ε, Opel, τη Vauxhall, τη Saab και ποια άλλη είναι. Αυτά είναι. Opel, Vauxhall, Saab. Αυτές οι τρεις. Ναι, η Volvo ανοίξει τη Ford. Λοιπόν, δεν μπορείτε να τους απαλλάξετε από την ευθύνη που έχει για αυτές τις θηγατρικές όποιος αυτή τη στιγμή δεσμεύεται εκ μέρους της Ευρώπης, ευκολύνει μόνο τη μητρική εταιρεία και το κάνει, κάνει την υπόθεση αυτή πιο ακριβή για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Χαίρομαι για το ότι καταφέραμε με τις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών να καταλήξουμε σε μία ξεκάθαρη συμφωνία για το ότι δεν υπάρχουν εδώ πέρα εθνικοί μονόδρομοι εθνική, εθνικές μεμονωμένες λύσεις θα οδηγήσουν στο ότι θα ε, βγει μια επιχείρηση η οποία δεν θα είναι οπωσδήποτε ανταγωνιστική και έτσι δεν βοηθάμε τους εργαζόμενους. Δεν τους βοηθάμε αν οι αποφάσεις ε, δεν λαμβάνονται με κριτήρια οικονομικά αλλά πολιτικά. και είναι ο κίνδυνος μετά πολύ μεγάλος της αποτυχίας. Κάναμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία με τις ε, κυβερνήσεις ότι ό,τι και αν συμβεί, εάν καταφέρουμε να σωθούν οι επιχειρήσεις και οι θέσεις ε, εργασίας και κυρίως γι' αυτό μιλάμε, θα γίνει αυτό με έναν τρόπο που θα ε, είναι σωστός οικονομικά Δεν έχει νόημα να δώσουμε δισεκατομμύρια για να σώσουμε μια επιχείρηση μόνο για μια εκλογική θητεία. Δεν είναι και υπεύθυνο αυτό. Αυτό το οποίο επίσης ε, κάναμε είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ε, μετατροπής αν θέλετε του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τοπίου σε ένα όχι μεταβιομηχανικό αλλά σε ένα διαφορετικό βιομηχανικό μέλλον. Χρειαζόμαστε πράγματι μια ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά θα έχει διαφορετική όψη από αυτή που είχε στο παρελθόν από την βιομηχανική επανάσταση και εδώ. Κάποια πράγματα, πράγματι, κύριε και κύριοι, δεν τα ολοκληρώσαμε. Γνωρίζετε πως το Κοινοβούλιο ασχολείται ακόμα με την πρόταση Κομισιόν για τα οικοδομικά υλικά, για το φαρμακευτικό πακέτο και θα έρθουν και άλλες ακόμα σημαντικές προτάσεις, οποίες δεν θα ήθελα να αναφέρω γιατί κατ' ουσία να αφορούν και το επόμενο Κοινοβούλιο. Ένα θα ήθελα να σας επισημάνω ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα και αφορά άμεσα την ε, εσωτερική αγορά Θα καταθέσουμε μεθαύριο μία πρόταση της ε, Κομισιόν για την καθυστέρηση και των ε, πληρωμών. Πρόκειται για μία πάρα πολύ σημαντική πρόταση, πολύ σημαντικότερη από όσο αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη και θα αντιμετωπίσει κυρίως ένα ε, ζήτημα ριζικά το οποίο για μένα είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο, δηλαδή το γεγονός ότι όλο και περισσότερο οι δημόσιοι φορείς είναι αυτοί οι οποίοι καθυστερούν τις πληρωμές. Και ξέρετε τι γίνεται. Ε, Μία μικρομεσαία επιχείρηση η οποία έχει, να λαμβάνει, έχει λαμβάνει αλλά θα εισπράξει σε 90 μέρες δεν θα επιζήσει αυτές τις 90 μέρες. Και πιστέψτε με χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες ε, θέσεις εργασίας κάθε χρόνο στην Ευρώπη γιατί χρεοκοπούν οι επιχειρήσεις λόγω των καθυριμένων πληρωμών. Και δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε αυτό από τον δημόσιο τομέα ο μέσος όρος πληρωμών από το δημόσιο ταμείο σε ε, και τέτοια είναι 120 μέρες. Και πάνω από αυτό. Οπότε θα έχουμε ριζική αναμόρφωση του σχετικού δικαίου και αν υπάρχει η λογική προσδοκία κάποιο ο οποίος έχει να λαμβάνει από το δημόσιο θα βλεωθεί εντός 30 ημερών. Και δεν θα επιτρέπεται να προκηρύξει κανείς διαγωνισμό χωρίς να έχει τα λεφτά στον προϋπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Και... Και οπωσδήποτε θα είναι πολύ έντονη εδώ πέρα η συζήτηση και θα ήθελα να, είναι, να σταθεί στο πλευρό μου εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας πω ένα νούμερο μόνο. Οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν 16% του συνολικού ΑΕΠ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ που αποτελούν δημόσιες προμήθειες. Εάν μιλάμε λοιπόν για αυτές πολύ μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμές, φαντάζεστε ποια είναι τα αποτελέσματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κυρίες μου και κύριοι, σε αυτά θα ήθελα να μείνω. Ε, τελειώνοντας ε, να πω το, το εξής. Αυτό το οποίο εκτίμησα εγώ πολύ ε, όσον αφορά την Επιτροπή σας είναι πως ε, κινηθήκατε διακομματικά και επικοδομητικά και με συνένεση και επικεντρωθήκατε στα, στα πράγματα και αποτέλεσε η συνεργασία μαζί σας ε, μία από τις πιο ευχάριστες πτυχές ε, της δουλειάς μου τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και γι' αυτό. Well, thank you very much, Commissioner. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής που είναι εδώ. Ε, θέλω να σας πω ότι είμαστε ρεαλιστές, ε, έχουμε πραγματιστική προσέγγιση. Ε, είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά διακυβευόμενα για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, τις θέσεις απασχόλησης, δεδομένης και της σημερινής κρίσης. Ε, είναι τα σχόλιά σας για την καλύτερη νομοθεσία. Εμείς ε, αυτό το θέμα το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Έχουμε χρησιμοποιήσει το 150% του προϋπολογισμού μας για μελέτες, ούτω ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνουμε να βασίζονται σε στοιχεία. Το μόνο θέμα που δημιουργεί πρόβλημα μερικές φορές στα κράτη-μέλη, και στην Κομισιόν, είναι ότι βρίσκουμε ότι οι μερικές ε, μελέτες επιπτώσεων δεν ευσταθούν. Εμείς θα συνεχίσουμε οπωσδήποτε να συνεργαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αλλιώς ε, αμαυρώνεται το όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάποιο χρόνο για ερωτήσεις. Νομίζω πως ναι, ναι, έχει και ο Επίτροπος. Το επόμενο θέμα είναι δικό μου και μπορώ να χρησιμοποιήσω λιγότερο χρόνο θα διαβάσω τον κατάλογο των ομιλητών. Um, Κινάμε με τον κύριο Χάρμπορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, όπως και εσείς, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Φερχόγγεν για τον τρόπο που συνεργάζεται με την Επιτροπή μας για την προθυμία του να έρχεται εδώ να μας επισκεφθεί. Αυτό που εκτίμησα ιδιαίτερα σήμερα το απόγευμα είναι ότι θέτει την εργασία μας μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων της οικονομίας και τις διάφορες ε, παραπλήσιες ε, πολιτικές. Τώρα που τελειώνει η θητεία του, θα ήθελα να μας συμβουλέψει για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Είναι τα πέντε πρώτα χρόνια της ε, Επιτροπής όπου ε, διαχωρίσαμε πολύ τις πρακτικές μας και τη δουλειά μας σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά για τα αγαθά και την εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες. Δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτό λειτουργεί. Νομίζω και σχολιάστε το ότι Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου η νομοθεσία για την εσωτερική αγορά είναι οριζόντια. Όλοι οι επίτροποι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή των νομοθετημάτων για την εσωτερική αγορά. Αν δούμε και την παράλληλη δουλειά που γίνεται ε, για το πακέτο αγαθών και υπηρεσιών που απαιτείται από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ενιαία σημεία επαφής για να ενημερώνουν τους φορείς την, ε, της οικονομίας τους για τη δυνατότητα πρόσβασή τους στην αγορά, νομίζω ότι η καινούργια επιτροπή θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό το θέμα. Επίσης, τις δημόσιες προμήθειες που επηρεάζουν πάρα πολύ και τα αγαθά και τις υπηρεσίες θα πρέπει να τις σκεφτούμε. και που μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην καινοτομία. Είναι στο τομέας αδιερεύνητο. Ε, καινοτομία και δημόσιε προμήθειε, δηλαδή. Τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ ενισχύεται και το επιχείρημά μου ότι υπάρχει σχετική έλλειψη συντονισμού στην ε, Επιτροπή. Δηλαδή, ε, η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης και κοινωνία της πληροφορία έχει ασχοληθεί με το θέμα δημοσίες προμήθεια, παύλα, καινοτομία. Εσείς θα μπορούσατε να έχετε πιο ανεξάρτητη άποψη ε, για το πώς εμεί ω Επιτροπή θα πρέπει να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και, το, και για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το προσεγγίσει. Αυτό ισχύει και για την ε, καλύτερη νομοθεσία. Νομίζω ότι οι υπηρεσίες σας λαμβάνουν πολύ στα σοβαρά το θέμα της καλύτερης νομοθεσίας. Αλλά δεν υπάρχει το ίδιο επίπεδο ποιότητας ε, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία και την εφαρμογή σε άλλες υπηρεσίες της ε, Επιτροπής. Και ο επόμενος Επίτροπος νομίζω θα πρέπει να πάρει αυτό το θέμα πολύ πιο σοβαρά καθώς και πρώτος του Κοινοβουλίου. Ε, ο οποίος άσκησε κριτική. Νομίζω ότι και εμείς πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά τις ευθύνες μας. Ίσως θα μπορούσατε να συμφωνήσετε μαζί μας και να πείτε ότι όλα τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου, που θα είναι και πολύ άριθμα, που θα εκλεγούν από τις εκλογές του Ιουνίου, όταν φτάσουν εδώ τον Ιούλιο, μαζί με τις ευρωπαϊκές ε, συνθήκες, θα πρέπει να έχουν και έναν οδηγό για την καλύτερη νομοθεσία. Ε, το έχω δει στο ίντερνετ, αλλά δεν έχω δει κανένα φυλάδιο για την καλύτερη νομοθεσία. Εν πάση περιπτώσει, κανένα φυλάδιο να έχει σταλεί στα μέλη του Κοινοβουλίου. Τι νόημα έχει να έχουμε καλύτερη νομοθεσία, να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση, αν δεν ενθαρρύνουμε τα μέλη του Κοινοβουλίου να το λαμβάνουν υπόψη αυτό το θέμα Νομίζω ότι τον απομείνοντα χρόνο που έχετε θα θέλατε να προωθήσετε αυτό το θέμα και ίσως να μιλήσετε και στα νέα μέλη για το πώς ε, θα μπορούσαν να καταστήσουν πραγματικά λειτουργική την καλύτερη νομοθεσία. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να τα πούμε μεταξύ μας. Είχατε συγκεκριμένη ευθύνη για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, κάτι πολύ σημαντικό. Το τελικό μου ερώτημα, το οποίο μπορεί να σας ενοχλήσει λίγο, είναι αν η ανταγωνιστικότητα είχε δείχτη 100 τον Ιούνιο του 2004 όταν ξεκινήσατε. Τώρα, πώς θα βαθμολογούσατε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πέντε χρόνια μετά, πέντε χρόνια μετά ε, την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Επίτροπου. Εντάξει, επειδή είναι τελευταία συνεδρίαση δεν θα είμαι τόσο αυστηρή στον χρόνο ομιλία. Η κυρία Βάιλερ. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ θα χαιρόμουν αν δείχνατε την ίδια επίκαια και σε μένα, που είναι η τελευταία συνεδρίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με της ομάδας μου τον κύριο Φερχόγγεν και για την ευθύτητα και την ακαιρεότητα που υπερασπίστηκε πάλι, πάντοτε την ε, ενιαία αγορά. Γνωρίζετε και θα το κρύψω ότι καμιά φορά διαφωνούσαμε, έτσι έχει η ζωή τι να κάνουμε. Ε, από την άλλη όμως ξεκαθαρίζεται πάντα και στην Επιτροπή μας εδώ αλλά και ε, δημόσια ότι η οικονομική πολιτική, η πολιτική της ενιαίας αγοράς δεν ισούται αυτόματα με τον άκρατο ε, φιλελευθερισμό και την ασυδοσία της αγοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν έρθω στις τρεις μου ευχές και επιθυμίες, θα ήθελα να αναφέρω δύο μικρά σημεία που είπατε κι εσείς. μιλήσατε για τις καθυστερήσεις πληρωμών και θα επιληφθείτε προσωπικά πριν αποχωρήσετε. Παρακαλώ και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να το πράξουν αυτό, γιατί σε ό,τι μας αφορά εμάς προσωπικά ως βουλευτές, υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Πολλές φορές εμείς προκαταβάλουμε ποσά για να μην περιμένουμε μικρές επιχειρήσεις. Και μερικές φορές περιμένουμε δύο με τρεις μήνες για τις πληρωμές που κανονικά ο στόχος είναι δύο με τρεις εβδομάδες. Μάλιστα, βλέπω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς, ε, το αναγνωρίσατε. Ξέρετε τι... Α, καλά που μπήκε και ο κύριος Φαπ τώρα. Επίσης μιλήσατε για τα ε, όπλα, για την νομοθεσία περί όπλων. Τουλάχιστον στη Γερμανία, ο τύπος ε, ε κατά σύμπτωση αυτό το έγραψε γιατί ένας επαρχιώτης πολιτικός από τη Βάδη Βουρτεμβέργη είπε, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, ε, ότι στο μέλλον, λες και ήταν αυτό επίτευγμα, ε, θα καταγράφονται όλα τα όπλα και μια συνάδελφος της Βουλής των Πρασίνων είπε ότι δεν είναι δικό σου επίτευγμα του επαρχιακού πολιτικού της Τσέντεου, της δεξιάς, αλλά της Ευρώπης. Έτσι και αλλιώς είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε, είτε το θέλετε είτε όχι. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα σημείο των καιρών και ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για ας πούμε εκτάκτους ελέγχους χωρίς προειδοποίηση όπως το ντόπινγκ ας πούμε σε ε, εκείνους που κατέχουν νόμιμα όπλα. Και τώρα κάνω τρεις ερωτήσεις. Ε, στην αρχή είπατε κάτι για τον προστατευτισμό, τον υπαρκτό ή τις απόπειρες και τους κανόνες που έχουμε και κατά πόσο αυτό αντιτίθεται στους κανόνες αυτούς. Εγώ δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για τη Γαλλία, αλλά διαβάζω πάντα ότι ε, η γαλλική κυβέρνηση και η γαλλική οικονομία προσπαθούν ό,τι κάνουν για να κινηθούν στο περιθώριο ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να προστατεύσουν τη χώρα τους υπάρχει αυτή η κουλτούρα του ρήνου, η λεγόμενη ο προστατευτισμό και δική μου χώρα δεν είναι τελείως αθώα εκεί. Αλλά πώς μπορούμε να βγαίνουμε στις χώρες μας και να λέμε τι να πούμε στους δικούς ψηφοφόρου όταν επιτρέπετε τα πάντα στους Γάλλους. Δεύτερον, ξέρω ότι δεν τονίζεται τόσο πολύ η κοινωνικότητα των εργαζομένων, employability, δηλαδή η απασχολησιμότητα. Το αναφέρετε με κάποιο τρόπο, νομίζω το επικρίνατε πολύ. Εγώ ζω σε μια περιφέρεια που είναι πάρα πολύ φτωχή από υποδομές και γνωρίζω εκατοντάδες εργαζομένους που ε, πρωί βράδυ έχουν πάνω από μία ώρα διαδρομή για να πάνε να δουλέψουν. Χιλιάδες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα βεβαίως και μετεκπαιδεύονται και αυτοί για να έχουν και πιο εύκολες συνθήκες, να μην χρειάζεται ε, να τους τρώει ο σιδηρόδρομος ή ο δρόμος κάθε μέρα όλες ολόκληρες. Και ένα τελευταίο είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση. Είπατε ότι... Δεν έχουμε αρκετή παιδεία και εκπαίδευση για το τι εστί επιχειρήν. Συμφωνώ. Και είναι πραγματικά ε, ε, πώς να το πω, πάρα ε, πολύ κακό, κακολέφριο να θέλουν όλοι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν ε, τονώνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, το επιχειρήν, δεν ενθαρρύνεται κτλ. Και τώρα και στο μέλλον φαντάζομαι χρειάζονται πολύ περισσότερες επαφές και θα έχετε εσείς και προς τη βιομηχανία και προς την ιδιωτική οικονομία. Θα παρακαλούσα να το έχετε αυτό υπόψη σας και ως επιθυμία και ως ευκή. Φέρουν και οι επιχειρήσεις ευθύνη σε αυτό. Και βέβαια τα θεσμικά όργανα, οι θεσμοί, κάνουν κατάρτιση, κάνουν εκπαίδευση, αλλά περισσότερο εμφανίζουν τα πράγματα μονομερώς. Για παράδειγμα, ότι ε, δεν, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, δεν χρειάζονται πάντα συνδικάτα, όχι. Ε, και αυτό ανήκει στην ε, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όχι να μαθαίνουμε στους άλλους πώς να είναι επιχειρηματίες, αλλά και ε, τη συνδικαλιστική κοινωνική δράση, τον κοινωνικό διάλογο. Παρακαλώ να το θέσετε αυτό υπόψη και των εργοδοτικών ε, οργανώσεων. Σας ευχαριστώ και πάλι από την πολιτική μου ομάδα και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Αγγελάκας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί πρέπει να φύγω να πάω να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή, αλλά θέλω να υποβάλω την ερώτηση. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη συνεργασία που είχαμε. Έκανε μία αναφορά στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Μιλήσατε κύριε Αντιπρόεδρε. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι αδύνατο να ανταγωνιστεί τις βιομηχανίες των τρίτων χωρών και αυτό που την διαφοροποιεί είναι η ποιότητα και η πρωτοτυπία. Είναι γνωστό ότι τρεις στις δέκα καινοτομίε μόνο δημιουργούνται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τουλάχιστον μόνο τρεις επιστήμονες από αυτούς που λέμε μυαλά παραμένουν στην Ευρώπη για να δραστηριοποιηθούν στον ερευνητικό τομέα. Θέλω να μας πείτε ποια πραγματικά πιστεύετε ότι είναι τα κίνητρα εκείνα που θα δημιουργήσουν ρεύμα επιστροφής ερευνητικών κέντρων στην Ευρώπη και ρεύμα επιστροφής επιστημόνων στην Ευρώπη. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να ακούσω την απάντησή σας, αλλά θα την πληροφορηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Mrs. Σας ευχαριστώ για τον απολογισμό τον οποίον κάνατε πράγματι είναι ευπρόσδεκτος. Νομίζω πως όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ πέρα συμφωνούν μαζί σας όταν λέτε πως ε, χρειαζόμαστε καλύτερη ρύθμιση. Π.χ. χρηματαγορές. Μπορεί όμως να διαφέρουμε όσον αφορά την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να πηγαίνει αυτή η καλύτερη ρύθμιση. Δηλαδή για κάποιους σημαίνει πως η καλύτερη ρύθμιση είναι η μη ρύθμιση. Το δε κοινοβούλιο ε, πάντα καταθέτει πολλές ε, τροπολογίες στις ε, προτάσεις της Κομισιόν, αλλά εάν δούμε και το τι έρχεται από πλευράς του, του 10 έχουμε τα εξής αποτελέσματα. Είτε ότι δεν υπάρχει ρύθμιση, είτε ότι οι κανόνες που υπάρχουν δεν είναι αρκετά σαφείς. Ε, και εσείς μας λέτε πως είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες που βάζει ορισμένες φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να μην καταλήξουν αυτά τα θέματα ενώπιον του ΔΕΚ, το οποίο τελικά θα είναι αυτό το οποίο θα αναγκαστεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Επίσης, ε, πρέπει να σας πω ότι η σημερινή κρίση μας αποδεικνύει ότι μερικές φορές και εμείς ε, κινηθήκαμε προς επικίνδυνες και αδικαιολόγητες ε, πολιτικές και οι χαμένοι ποιοι είναι, οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμη και εσείς το είπατε, Επίτροπε. Όταν μία επιχείρηση έχει 5.000 εργαζόμενους, το κράτος έχει σχεδόν την υποχρέωση να παρέμβει για να σώσει την επιχείρηση. Δυστυχώς, παρά τις δηλώσεις καλών προθέσεων, το κράτος δεν παρεμβαίνει όταν μια επιχείρηση είναι πολύ μικρή και έχει 5 εργαζομένους. Τότε τη θυσιάζει. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε τα δεδομένα λαμβάνοντα υπόψη την πραγματικότητα. Να σα κάνω μια άμεση ερώτηση. Πρόσφατα υπήρξαν πολλέ νομοθετικέ πρωτοβουλίε για τι επιχειρήσει και την οικονομική πολιτική. Και εσείς ο ίδιος τις προωθήσατε. Από εσά ξεκίνησαν πολλές από αυτέ τις πρωτοβουλίες. Υπάρχουν επίσης πρωτοβουλίες για την προστασία του καταναλωτή και για την κοινωνική πολιτική. Θα ήθελα να μάθω πώς μπορούμε να συνδέσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, τις νομοθετικές, για την επιχείρηση και τους καταναλωτές και την κοινωνική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Τι αποφάσεις έχει πάρει η Κομισιόν. Φαντάζομαι ότι οι αποφάσεις που παίρνετε ούτως ή άλλως είναι συνενετικές. Επομένως ε, και εσείς ε, συμμετείχατε στην προώθηση άλλων πολιτικών, όχι μόνο αυτές που αφορούν το δικό σας τομέα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε συγκεκριμένα τι έκανε η Κομισιόν. Ο επόμενος ομίλητης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε που μας επιτρέψατε να ακούσουμε αυτόν τον απολογισμό, ο οποίος είναι πολύ απαραίτητος, πολύ χρήσιμος. Δύο παρατηρήσεις και μία ερώτηση. Πρώτον, πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση του προστατευτισμού κάποιων χωρών όπως η Γαλλία, είπαν ορισμένοι συνάδελφοι. Θα ήθελα στην επόμενη νομοθετική θητεία να ασχοληθούμε περισσότερο με την κοινωνική προτίμηση, γιατί το νομοθετήν σημαίνει και μείωση του προστατευτισμού υπέρ των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα εδώ μεταξύ κάποιων εναρμονήσεων που μας επιτρέπουν αυτή την κοινοτική πρόταση και μιας εσωτερικής έτσι, και εντελώς προστατευτικής εθνικής πολιτικής σε ορισμένε χώρες. Έτσι. Δεύτερον, σε ορισμένε χώρες η κρίση επιταχύνει τα προβλήματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδυναμώνεται, ενώ άλλες περιφερειακές δυνάμεις όπως η Κίνα ε, ε, γίνονται πολύ πιο επιθετικές, πολύ πιο δυνατές. Πολλοί από εμά κρούσαμε τον κόδωνα. Πιστεύουμε ότι μια καλύτερη εσωτερική αγορά επιτρέπουμε την ενδυνάμωση με σκοπό την δημιουργία εταιρικών σχέσεων για να χρησιμοποιήσουμε την παγκοσμιοποίηση παρά να την υφιστάμεθα. Σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως έδειξαν πολλές οδηγίες, Αν απλουστεύσουμε την νομοθεσία υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, τους δίνουμε χώρο να αναπνεύσουν, ε, ώστε να ανταγωνιστούν και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα λοιπόν. Η Επιτροπή μας μαζί με την Ευρωπαϊκή Πολιτική θα πρέπει να προωθήσει πολύ πιο στεναρές πολιτικές. Όχι αυστηρές, όχι σκληρές αλλά στεναρές, ε, μαζί με τις τρίτες χώρες. Κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Πολιτικές μαζί με τις τρίτες χώρες. Και ένα τελευταίο. Πολύ συχνά ξεχνάμε ότι η απουσία εμπιστοσύνης που αυτές οι επιχειρήσεις υφίστανται, γιατί οι καταναλωτές δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά, θα μπορούσε να καλυφθεί από ένα εργαλείο που νομίζω ότι είναι εκ των Είναι η προστασία του καταναλωτή, ακριβώς. Να αντιπαρατεθούν οι προστατευτικές πολιτικές απέναντι στις πολιτικές προστασίας του καταναλωτή. Αυτό το είδαμε με πολλά θέματα, με πολλά κείμενα, με πολλά νομοθετήματα συχνά η στάση μας ήταν αποπροσανατολισμένη. Μερικές φορές ψηφίσαμε υπέρ των κειμένων, μερικές φορές ψηφίσαμε κατά. Νομίζω ότι ο φάρος που θα μας κατευθύνει θα είναι η προστασία του καταναλωτή. Αυτό μπορεί να, είναι, μπορεί να υπάρξει και ένα εργαλείο έτσι, ρύθμισης. Γιατί όταν υπάρχει εμπιστοσύνη του καταναλωτή, υπάρχει ανάκαμψη της ε, κατανάλωσης και επομένως ε, έχουμε πιο εύρωστες επιχειρήσεις. Το είπε και στην αδελφός μου. Όσο υπάρχουν ε, θέματα που καταφεύγουν στο ΔΕΚ, όσο περισσότερα είναι τα θέματα λοιπόν που πρέπει να τα διευθετήσει το ΔΕΚ, τόσο λιγότερο πιστικές είναι οι μας. Ελπίζω αυτό να διορθωθεί στην επόμενη θητεία. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τώρα και να ολοκληρώσετε κύριε Επίτροπε. Τέθηκε το θέμα του ελέγχου της πρόσβασης στα όπλα από σας Επίτροπε και από κάποιους συναδέλφους. το... Συχνά είπαμε ότι, το είπαν και συνάδελφοι, ότι όταν πάει κάτι καλά το καρπώνται τα κράτη-μέλη. Όταν, όταν κάτι άσχημα, κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε ένα κράτος μέλος που ζητούσε πιο αδύναμη νομοθεσία ε, και όμως όταν ψηφίσαμε την ε, σχετική κοινοτική νομοθεσία ε, απήχε ε, παραπέμποντας τη δική του εσωτερική νομοθεσία. Όλα αυτά τα θέματα ουσιαστικά πάντα είναι για τους πολίτες μας, έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που ακούσαμε, πάρα πολλά θέματα που τέθηκαν. Θα ήθελα να απαντήσετε και να κλείσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με τις παρατηρήσεις ε, του φίλου μου του Μάλκομ Χάρμπορ. Δύσκολο ερώτημα το εάν ε, η Επιτροπή πρέπει να ασχολείται με ζητήματα εσωτερικής αγοράς ε, ε, αγαθών κτλ. Αυτό σχετίζεται με την εσωτερική διάρθρωση του οργανισμού μας το συζήτησα αυτό και με κάποιον πολιτικό από την περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και απάντησα εγώ ως εξής. Εγώ θεωρώ πως καλό είναι να συγκεντρωθούν ε, σε ένα σημείο οι αρμοδιότητες της εσωτερικής αγοράς γιατί υπάρχουν τόσο πολλές επικαλύψεις. Είναι τόσο τεχνητοί οι διαχωρισμοί που για μένα είναι ζήτημα πολιτικού χειρισμού και μπορεί να είναι πολύ μεγάλη η διαφορά του με ποια φιλοσοφία θα προσεγγίσει κανείς το, το ζήτημα της ρύθμισης μιας μεγάλης αγοράς με τη φιλοσοφία της ε, κοινωνικής οικονομίας αγοράς ε, ή ε, παραδείγματος χάρη με μια ακραία προσέγγιση της αγοράς. Εκεί πέρα οδηγούμαστε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα και προσεγγίσεις. Εγώ νομίζω πως ε, καλό θα είναι κατά τη διαμόρφωση αυτής της ε, αγοράς να υπάρχει ένας ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την ε, πολιτική της εσωτερικής αγοράς. Τώρα για την καινοτομία. Για αυτό το οποίο είπε ο Μάλκομ. Συμφωνώ. Πράγματι παρά το ότι η Κομισιόν είναι έτσι οργανωμένη ώστε να μην υπάρχει ποτέ έλλειψη τυπικής, ε, τυπικού συντονισμού ή γίνονται τόσο πολλές ε, συνεδριάσεις αλλά εμείς ως πολιτικοί γνωρίζουμε πως η φυσιολογική, η φυσιολογικό συντονισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό ο αποτελεσματικό συντονισμός από τον πολιτικό συντονισμό. Και αντιλαμβάνεστε βεβαίως πως όταν μιλάμε για τον εσωτερικό συντονισμό υπηρεσιών της Κομισιόν, ε, το πώς θα γίνει αυτό με τους το, πολλούς διαφορετικούς ε, παίκτες, αν θέλετε, στον τομέα της καινοτομίας, γιατί έχουμε πολλούς φορείς, ε, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς κτλ. κτλ. Οπότε μία προσπάθεια της Κομισιόν να επιτύχει μια ριζοσπαστική αλλαγή ήταν αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας το Ευρωπαϊκό Πολυτεχνείο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα αυτής της ε, πρωτοβουλίας, γιατί είναι ακόμα στην αρχή. Ελπίζω να μην σας δημιουργήσω την εντύπωση ότι είμαι απογοητευμένος από την θητεία μου, αλλά το πόσο αργά κινούνται ορισμένα πράγματα στην Ευρώπη είναι, ε, είναι πραγματικά απογοητευτικό και Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Όμως πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού θα, γίνουμε, θα γίνουν κάποιες στρατηγικές σκέψεις για τη μεσαλλοντική ευρωπαϊκή πολιτική της ε, καινοτομίας. Αν θέλετε έτσι για να βοηθήσουν την επόμενη Κομισιόν και το επόμενο Κοινοβούλιο με βάση τις εμπειρίες που έχω κάνει, που έχω ζήσει εγώ. Οπότε θα έχουμε αυτή τη μεγάλη στρατηγική ανακοίνωση της Κομισιόν πριν από τις διακοπές. Σας ευχαριστώ επίσης πολύ για την διαρκή στήριξη την οποία μου έδειξε αυτό το κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας ε, όσον αφορά το έργο αυτό της καλύτερης νομοθεσίας και ε, μπορώ να ελπίζω μόνο πως θα συνεχιστεί κάτι τέτοιο και πως όλοι είναι διατεθειμένοι να μάθουν ε, και τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, κύλησαν όλα τέλεια, είχαμε πρόοδους, αλλά όπως πάντα όταν κανείς είναι πρωτοπόρος η πρόοδος δεν είναι πλήρης. Μάλκομ, αν μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, όταν ο Καρλ Μπέντς εφήβρε το, το αυτοκίνητο, ο γιατί ο Καρλ Μπέντς ήταν και όχι ο, οι Αμερικανοί, όπως ε, ισχυρίζονται πρόσφατα, ήταν μια τεράστια τεχνολογική καινοτομία. Αν βλέπαμε σήμερα αυτό το αυτοκίνητο, ε, ε, είναι, είναι πραγματικά συγκινητικό, αλλά δεν θα ήθελα εγώ να το, να το οδηγήσω, καταλαβαίνετε, να, να έχω αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή όταν κάποιος ξεκινάει μια διαδικασία, η οποία είναι πολύ μακροπρόθεσμη, τότε εντάξει, εάν κοιτάει τις ίδιες του τις προσπάθειες μετά εκ των υστέρων, μοιάζουν μικροί, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι τα πρώτα βήματα είναι τα δυσκολότερα και τα σημαντικότερα. Εντάξει, δεν έχω ψευδοστήσεις. Είμαστε ακόμα στην αρχή λοιπόν κι εμείς. Ναι, και κάτι ακόμα ρώτησε ο Μάλκομ. Εάν ε, θέταμε έναν ε, δίκτυ και το 2004 ήμασταν στο 100 ας πούμε, σήμερα που έχουμε φτάσει σήμερα ας πούμε, σε σχέση με τις είπα ή με άλλη. Τέλος και με τα δύο θα δούμε. Όσον αφορά την παραγωγικότητα, κάπου μεταξύ 108 και 110 θα έλεγα ότι θα, θα ήταν σήμερα ο δείκτης. Εντάξει, καλό αποτέλεσμα για μερικά χρονάκια μόνο. χοντρικά αυτά, Μάλκομ, έτσι. Αλλά ευχαρίστως να βάλω τους εικονομέτρες ε, να το δουν το, το ζήτημα και να σου δώσουν πιο ακριβείς αριθμούς. Μπάρμπαρα Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ για τα φιλικά σου λόγια και για την στήριξη. Θέλω να τονίσω το εξής. Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ έτσι, ριζοσπαστικός αγοράς. Εγώ ήμουν θα έλεγα του καπιταλισμού του Ρήνου. Δηλαδή αποδέχομαι πλήρως τα, τα συνδικάτα. Είναι καλά, καλό για τις επιχειρήσεις το να υπάρχουν συνδικάτα που λειτουργούν. Το αναγνωρίζω είναι επίσης υπέρ του οικονομικού μοντέλου με το οποίο εγώ μεγάλωσα και ήταν ε, επιτυχημένο. Ε, ήταν μάλιστα το πιο επιτυχημένο στην Ευρώπη κάποτε το, το, οικονομι, το μοντέλο της ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και βέβαια σήμερα πρέπει να το δούμε πάντα σε συνάρτηση με την οικολογία, τώρα πια δεν συνδέεται μόνο με το εισόδημα, αλλά και αλληλεγγύη με τις επόμενες γενιές. Οπότε το μοντέλο της οικονομίας αγοράς το οποίο εγώ πιστεύω είναι ένα μοντέλο το οποίο λαμβάνει υπόψη και έχει ευθύνες κοινωνικές και οικονομικές, πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Και δεν ε, θα συμφωνούσα με το ότι όσον αφορά την καλύτερη νομοθεσία η φιλοσοφία είναι καλύτερα ή να μην κάνουμε τίποτα τότε. Αυτό ως απάντηση στην κυρία Κρετού. Η πολιτική αυτή δεν εξισώνεται με την απορρίθμιση, ε, την Απορρίπτω αυτή την προσέγγιση. Δεν μιλάμε για απορρίθμιση. Μιλάμε για το να επιτύχουμε κάποιες προδιαγραφές με τον απλούστερο και καλύτερο τρόπο και με το να μην έχουμε άσκοπο κόστος. Και το βάρος είναι στη λέξη άσκοπο. Υπάρχει κόστος και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Επίσης ευχαριστώ την Μπάρμπαρα για αυτό που με επενθύμησε για το δίκαιο των όπλων. Εντάξει, γνωρίζω πως εγώ δέχομαι τις ερωτήσεις, αλλά εφόσον πρόκειται περί Γερμανίδας βουλευτού, θα ήθελα να πω πως πόσο είναι δυνατόν όταν κάποιος ανήκει σε σκοπευτικό σύλλογο να έχει 24 όπλα στο, στο σπίτι του. Πώς θα προστατεύσουμε έτσι τους, τους συμπολίπους όταν δίνονται αυτές οι ελευθερίες στους Δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό έτσι. Είναι μια σειρά λοιπόν ερωτημάτων που πρέπει να τεθούν. Τώρα για την κυρία Βάιλερ, προστατευτισμό στη Γαλλία. Ξέρω ότι η Γαλλία πάντα έχει αυτή την υποψία να επικρεμάται από πάνω το κεφάλι της. Κοιτάξτε, να σας το πω έτσι. Ε, τα εργαλεία και οι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής επαρκούν και σε μεγάλα με κράτη-μέλη να τα αναγκάζουν να τηρούν τους κανόνες. Ε, το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι τα μεγάλα κράτη δεν στριμώχνονται. Η κυρία Νέλη Κρούσο όμως που είναι αρμόδια εδώ για την πολιτική ανταγωνισμού είναι τέτοια ε, ώστε όσο περισσότερο προσπαθεί να την πιέσει ένας αρχηγός κράτους και κυβέρνησης, τόσο λιγότερο θα ενδώσει αυτή. Μπορείτε να είστε βέβαιοι αυτό, έτσι είναι ο χαρακτήρας της. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ σταθερή πραγματικά αυτή η εταιρική μας σχέση. Γιατί από την αρχή εγώ κατάλαβα και ξέρω ότι ε, η ευημερία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εταιριών εξαρτάται πραγματικά από την ε, πολιτική του ανταγωνισμού. Μια που επενώ την Έλλη Κρούς, να συνεχίσω. Πέτυχε μια νέα αφετηρία, μια νέα αρχή στην καταπελώμηση των καρτέλ και την υποστηρίζω πλήρως. Ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια και δώσαμε, βάλαμε τα μεγαλύτερα πρόστιμα έχουμε επιβάλει στα καρτέλ ε, σε αυτή τη θητεία και ποτέ δεν θα έχουν προβλήματα μαζί μου, είπε εκείνη ε, που ε, φωνάζουν ε, να θέλουν κανόνες ανταγωνισμού υγιής και καλούς, αλλά θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι ίδιοι κάνουν καρτέλ στις πλάτες και εις βάρος των καταναλωτών. Και το πράττει κιόλα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση εδώ που υποτίθεται ήθελε η Γαλλία να δώσει ενισχύσει στην αυτοκινητοβιομηχανία και αυτό να συνδέεται με μια ρήτρα που να λέει να αγοράζουν ε, αυτοκίνητα στη Γαλλία. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, δεν συνδέθηκε. Αφήστε που κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο. Διότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι πανευρωπαϊκή και πολλά εξαρτήματα ε, που χρειάζονται για ένα αυτοκίνητο το οποίο μοντάρεται, συναρμολογείται στη Γαλλία, δεν παράγονται στη Γαλλία, δεν μπορείτε να τα βρείτε καν. Γιατί οι προμηθευτές είναι πάρα πάρα πολύ εξειδικευμένοι και διασπαρτοί σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, για τους εργαζομένους ήταν ε, μάλλον παρεξήγηση, μάλλον που γερμανικά μιλάω, βρε παιδιά. Δεν υπάρχουν για κινητικότητα εργαζομένα. Δεν μίλησα καθόλου για την κινητικότητα. Είπα για ελαστικότητα, ευελιξία, δηλαδή προσαρμοστικότητα στην κατάσταση. Όχι σε, νέ, σε νέους χώρους που εργάζονται ή ζούνε, αλλά προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις, όχι στη μετακόμιση. Αυτό εννοούσα. Και σε ό,τι αφορά την εταιρική ευθύνη, ε, μίλησα εκτενώς για την κοινωνική εταιρική ευθύνη Corporate Social Responsibility λέγεται αυτό, και είναι απολύτως αναπόσπαστο τμήμα πολιτικής ευρωπαϊκής επιχειρήσεων η κοινωνική ευθύνη και η κοινωνική εταιρική ευθύνη να μην θεωρείται ως ένα πάρεργο ε, δημοσίων σχέσεων ε, όπου έχει την πολυτέλεια εταιρεία να την κάνει όταν πάνε καλά οι δουλειές της, αλλά αποτελεί πραγματικά ένα απόσπαστο κομμάτι και θα πρέπει να είναι και στόχος της επιχείρησης. Οι εταιρείε λοιπόν που έχουν ε, καλό απολογισμό σε αυτό τον κλάδο, κανονικά είναι και οι πιο επιτυχημένες. Ο κύριος Αγγελάκας ζήτησε να τον ενημερώσουμε γραπτός πράγμα που θα πράξουμε κιόλα για την έρευνα ε, και πώς θα την ξαναφέρουμε πίσω στην Ευρώπη και την επιστήμη. Μα η απάντηση είναι ε, απλή. Να δημιουργήσουμε τις υλικές προϋποθέσεις και να τις βελτιώσουμε. Βέβαια, εδώ δεν εννοώ κυρίως το εισόδημα. Μιλάω πάρα πολύ με ερευνητέ και με επιστημονε που πήγαν στην Αμερική. Δεν πήγαν στην Αμερική γιατί θα βγάλουν πολλά λεφτά πιο γρήγορα, αλλά πήγαν κυρίω στην Αμερική γιατί οι συνθήκε εργασία είναι εκεί καλύτερε. καλύτερες. Γιατί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερε δαπάνε. Γιατί είναι πολύ πιο ελαστική, είναι πολύ πιο καλή. Ε, Κάποιο που είναι ερευνητή και έχει μια καλή ιδέα, βρίσκει και έναν άνθρωπο που να τον βοηθήσει να την κάνει πράξη. Ε, στην Ευρώπη σε πολλέ περιπτώσει αυτό δεν ισχύει. Είσαι ερευνητής σε ένα Ινστιτούτο, έχεις μια φανή ιδέα και μπορεί ε, δεχομένω η ιδέα αυτή να κολλήσει κάπου στην υπηρεσία και να του πούνε για ξανά έλα ε, ε, όταν θα έχεις δημοσιεύσει 25 έγγραφα και όταν θα έχεις κάνει και καμιά σοβαρή δουλειά. Ε, όχι, στην Αμερική αμέσως ενθαρρύνεται η καλή ιδέα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος, πιστεύω. Για την κυρία Κρέτσου είχα απαντήσει για την καλύτερη νομοθεσία. Αυτό δεν είναι απορρίθμιση καθόλου. Όπως λέει το όνομα, είναι ε, αύξηση της ποιότητας. Τώρα δεν μίλησα για τα άλλα σημεία, αλλά για μία μόνο παράγραφο, για να αποφύγουμε το άσκοπο γραφειοκρατικό κόστος. Τα άλλα σημεία που αφορούν τη μελέτη σκοτπιμότητα, επιπτώσεων και το evaluation και τις εκτιμήσεις, τις ανάγκες, διαβούλευσης. Όλα αυτά δεν τα ανέφερα, ανήκουν όμως στο συνολικό πακέτο και στο συνολικό σχέδιο. Και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ακολουθήσουμε τη γραμμή αυτή. Ο σωστός δρόμος δεν είναι η απορρίθμιση, αλλά οι σωστοί κανόνες, οι καλοί κανόνες, όχι ε, η απεμπόληση. Το έχω επανειλημμένα τονίσει γιατί χρειάζεται κατά τη γνώμη μου ε, κανόνιση αγορά. Άλλη ερώτηση. Ε, κοινωνική πολιτική, προστασία των καταναλωτών κλπ. και σύνδεση με αυτά. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όντως είναι πάντα συνεκτική. Γίνονται προτάσεις. Ποτέ δεν είναι αυτές προτάσεις με μονομένου επιτρόπου. Είναι πάντα ε, προτάσεις του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις κυρίας Κούνεβα, για παράδειγμα, για την προστασία των καταναλωτών, είναι κάτι και το οποίο και εγώ προάγω και υποστηρίζω, όπως άλλωστε και η κυρία Κούνεβα της δικές μου. Γι' αυτό είναι και συλλογικό το σώμα. Ε, αυτή την έννοια έχει ένα τέτοιο σώμα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια συλλογικότητα. Έτσι ώστε να συνδέονται και να υπάρχει συνοχή και συνάφεια. Βέβαια το παραδέχομαι, δεν το πετυχαίνουμε πάντα αυτό. Πάντως, ε, όλο και πιο συχνά. Συμφωνώ με όλες οι επικυριανέρεις, ε, ιδιαίτερα για το ρόλο των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων. Να σας πω κάτι για την παρατήρησή σας για τις τρίτες χώρες μόνο από ό,τι φαίνεται έχετε την εντύπωση ότι δεν συνεργαζόμαστε πάρα πολύ προς το σκοπό αυτό. Τώρα θα μπορούσα να σας καλέσω να προσπαθήσω να ε, δούμε τι γίνεται στην πράξη και θα καταλήγαμε και ίδιο στο συμπέρασμα ότι το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε αρκετό διάλογο, φόρα, συναντήσεις, συνεργασία και συνόδους κορυφής και ανακοινοθέντα. Πληθώρα τέτοιων έχουμε και πληθώρα επισκέψεων. Όλο και περισσότερο σκοτεινιάζει ο ουρανός στην Ευρώπη από αεροπλάνα που πετάνε. Ε, και είναι εκπρόσωποι άλλων κρατών και διοικήσεων που έρχονται εδώ να συζητήσουν μαζί μας και τούμπαλε. Αυτό που επέκνα εγώ δεν ήταν το γεγονός ότι δεν έχουμε επαφές με τις τρίτες χώρες, αλλά ότι ουσιαστικά βγαίνουν πάρα πολύ λίγα στην πράξη από τις επαφές αυτές. Με ξέρεις τις ΗΠΑ. Τώρα είναι και δημόσια συζήτηση. Δεν θέλω να δημιουργήσω διπλωματικές ε, δυσκολίες, αλλά υπάρχει μια σημαντική χώρα με την οποία κάθε χρόνο ανανεώνουμε τις συμφωνίες μας, ότι τα εμπόδια σε υπηρεσίες και στο εμπόριο με αγαθά και με κεφάλαια και τα λοιπά θέλουμε να τα εγκαταλείψουμε, αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν άλλαξε τίποτα, ούτε ένας κανόνας στην έλογο χώρα για να υλοποιηθούν όλα αυτά που μαζί αποφασίζουμε. Έτσι, το πρόβλημα λοιπόν για μένα δεν είναι τόσο πολύ στη δική μας πλευρά. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε βήματα, αλλά οι εταίροι μας και οι μεγάλες περιφέρειες αυτές και σημαντικές θεωρούν ότι θα πρέπει να ισχύουν άλλοι κανόνες γιατί έχουν ε, καθυστέρηση και θα πρέπει να την καλύψουν. Και για την προστασία των καταναλωτών τελευταίο, η συνοχή και η συνάφεια της πολιτικής που σας είπα προηγουμένως και η συνέχεια. Πώς ε, προκύπτουν καν οι ε, προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν συζητούμε μόνο για τα δικαιώματα των καταναλωτών εκεί, αλλά τα λαμβάνουμε πλήρως υπόψη και η κυρία Κούνεβα, την οποία γνωρίζετε όλοι, ε, έχει επιβολή. Δεν, ε, είναι άψογη ε, η λειτουργία της υπηρεσίας. Έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί το αντίθετο στην Ευρώπη. Και εδώ στην Επιτροπή σας. τα γνωρίζετε αυτά πάρα πολύ καλά. Διότι με τμήμα των οδηγιών που μαζί έχουμε ε, αποφασίσει και τον κανονισμό αφορά την ασφάλεια προϊόντων. Και προς όφελος ποιον τα ζητάμε όλα αυτά, των καταναλωτών. Ανδρών και γυναικών. Πάντως είμαι πάντα πρόθυμος να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για βελτιώσεις και όπου χωρούν αυτές να γίνουν. Βασικός κυρίαρχος στην αγορά είναι ο καταναλωτής ή θα έπρεπε να είναι. Ή θα έπρεπε, εν πάση λέγω. Και εμείς θα έπρεπε να κάνουμε μια πολιτική που να επιτρέπει στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί αυτό το προνόμιο και να το αξιοποιεί. Αυτό είναι και σημαντικό και χρήσιμο. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένας καταναλωτής ε, ενημερωμένος ε, που να μην παραπλανάται. που να διαθέτει και να χρησιμοποιεί ε, τις πληροφορίες που υπάρχουν το συντομότερο. Όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάντα θα βρίσκουν τη δική μου υποστήριξη. Κύριε Πρόεδρε, αυτά. Προσπάθησα να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σας. Τι άλλο να σας πω τώρα. Αυτά. Ολοκληρώνεται εδώ η συνεργασία μας και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Ως Επιτροπή θα ήθελα να σας ευχηθώ και προσωπικά και εξ ονόματος Επιτροπής ε, καλή τύχη. Φαντάζομαι ότι θα σας ξαναδούμε γιατί ούτως ή άλλως τα ταλέντα δεν θα χαθούν. Θα ασχολήσετε και στο μέλλον με, την, ε, με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ευχαριστώ και ευχαριστώ Επίτροπε. Θα προσπαθήσω να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Όσοι δεν ήσασταν εδώ από την αρχή, χάσαμε περίπου 20 με 25 λεπτά στην αρχή λόγω τεχνικών προβλημάτων με τη διερμηνία. Γι' αυτό καθυστερήσαμε λιγάκι. Τι προτείνω λοιπόν τώρα για το επόμενο σημείο που είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών. Να σας ε, ενημερώσω πολύ σύντομα ε, το τι συνέβη ε, στο Στρασβούργο στην ομάδα εργασίας και να σας ενημερώσω για ό,τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα και συνεχεία να περάσουμε στο καλεσμένο μας, ο οποίος θα μας μιλήσει για το σχέδιο πυρασφάλισης των πνευμαδοχείων. Στους καλεσμένους μας μάλλον, εμπειρογνώμονες. Εγώ λοιπόν δεν θα ξοδέψω πολύ χρόνο. Ευχαριστώ τους συντονιστές που παρέστησαν στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας στο Στρασβούργο. Συζητήσαμε ένα σχέδιο εγγράφου. Γιατί θα θυμάστε ότι οι συντονιστές είχαν πάρει μια πολιτική απόφαση ότι δεν θα κάνουμε πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο, ότι θα εκπονήσουμε ένα ενημερωτικό έγγραφο εργασίας. Ελήφθη απόφαση επίσης να υποβάλουμε ε, στην Επίτροπο Κούνεβα ε, μία προφορική ερώτηση, καθώς και μία απόφαση για μία άλλη προφορική ερώτηση που θα βασίζεται στα όσα αναφέρει το έγγραφο εργασίας. Τα μέλη της ομάδας εργασίας συζήτησαν τη δομή αυτού του εγγράφου, που είναι νομίζω αρκετά απλή και ουσιαστικά παρουσιάζει, θα σας μοιραστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί μέχρι τότε θα την ολοκληρώσουμε αυτή την έκθεση. Ουσιαστικά εξετάζει την πρόταση της Κομισιόν, τους στόχους της, εξετάζει με λεπτομέρειες κάποια βασικά στοιχεία ε, που αφορούν τη μελέτη επιπτώσεων, θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας της πρότασης. Εν συνεχεία, υπησύλθαμε σε κάποιες λεπτομέρειες της ε, πρότασης. Μην ξεχνάτε την ακρόαση που είχαμε διοργανώσει και την online διαβούλευση ε, όπου λάβαμε αρκετέ απαντήσεις, οι οποίες μας βοήθησαν πάρα πολύ και τις λάβαμε υπόψη για να συντάξουμε αυτό το έγγραφο εργασίας. Στο έγγραφο εργασίας εξετάζουμε το επίπεδο εναρμόνισης, το αν υπάρχει πλήρης εναρμόνισης, ε, το αν υπάρχει εστιασμένη εναρμόνιση ή αν θα πρέπει να υπάρξει εστιασμένη εναρμόνιση. Κάτι που, κάτι που είπαν πολλές ε, οργανώσεις καταναλωτών είναι ότι θα, προτιμούσαν μία ελάχιστη εναρμόνιση. Εν συνεχεία, το πεδίο της πρότασης, το πεδίο εφαρμογής της πρότασης, ακούσαμε κάποιες επικρίσεις στην ακρόαση και στη διαβούλευση online, ε, γιατί υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Εν συνεχεία μπήκαμε σε όλες τις λεπτομέρειες της πρότασης και θα θέλαμε να κλείνει αυτό το έγγραφο εργασίας ε, εξετάζοντας περιληπτικά τις υπόλοιπες εναλλακτικέ που έχουμε, που ακούστηκαν στην ακρόαση και στη διαβούλευση. Ξέρετε ότι υπάρχουν και εναλλακτικέ προτάσεις πέρα από την πρόταση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συντονιστέ είπαν ότι θα πρέπει ε, στο έγγραφο εργασία να παρουσιάζονται αυτές οι εναλλακτικέ λύσει χωρί να δεσμευόμαστε ε, υπέρ μία ή άλλη εναλλακτική λύσης όλα, το κείμενο αυτό θέλει να αντικατοπτρίζει όλες τις δυνατότητες. Η τελική απόφαση τώρα θα είναι έργο της νέας Επιτροπής. Εκεί θα, εκείνη θα ασχοληθεί με την πρώτη ανάγνωση, με τη δεύτερη ανάγνωση. Το άλλο θέμα είναι ότι ζητήσαμε από την Κομισιόν να προβεί σε περιττέρω ανάλυση γύρω από τις ανησυχίες ε, της πλήρους εναρμόνισης, τι σημαίνει αυτό και τι επιπτώσεις θα έχει στη, στους καταναλωτές. Θα θέλαμε η Κομισιόν να ξεκαθαρίσει τη σχέση μεταξύ της προσέγγισης της πλήρους εναρμόνισης και των δυνατοτήτων που μας δίνει η εθνική νομοθεσία στα πλαίσια του εταιρικού δικαίου. Η Κομισιόν, όπως είπαμε και στην ακρόαση και στη διαβούλευση, θα θέλαμε να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για τις, τα θετικά και τα αρνητικά των διαφόρων αλλακτικών λύσεων. Και μια και δεν θα γίνει η πρώτη ανάγνωση το Μάιο, έχουμε περισσότερο χρόνο για να μπούμε σε λεπτομέρειες. Μπορεί οι ενδιαφερόμενοι, οι stakeholders, ε, στα πλαίσια ενός διαλόγου μεταξύ των εθνικών ε, οργανώσεων καταναλωτών να καταλήξουν σε κάποια δέσμη δικαιωμάτων καταναλωτών που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Θα θέλαμε να βρούμε μια προσέγγιση η οποία να είναι πρακτική και ρεαλιστική και όπως είπαμε ήδη δεν θα υποδυναμητίζει τα σημερινά δικαιώματα των καταναλωτών ή θα δίνει στους καταναλωτές το, την εντύπωση ότι έχουν λιγότερα δικαιώματα. Και βεβαίως ε, θα εξασφαλίζει πρόσβαση στις επιχειρήσεις στις 27 εθνικές αγορές. Αυτή είναι η βασική στόχη της Επιτροπής μας που θέλουμε να προωθήσουμε την ελεύθερη αγορά την εσωτερική αγορά, αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών, να προωθήσουμε επίσης την παροχή υπηρεσιών και αγαθών στα εσωτερικά σύνορα. Αυτό το έγγραφο θα μοιραστεί σε όλους τους βουλευτές της Επιτροπής, όχι μόνο στους συντονιστές. Και εν συνεχεία οι πολιτικές ομάδες θα λάβουν μια απόφαση σε ό,τι αφορά την προφορική ερώτηση και το ακριβές περιεχόμενό της. Η Επίτροπος Κούνεβα έχει δηλώσει ήδη την προθυμία της να απαντήσει στην προφορική ερώτηση στην τελική ολομέλεια του σημερινού Κοινοβουλίου. Διάφορα μέλη, διάφοροι βουλευτές, ο κύριος, ο Χάρμπορ, είπε ότι θα πρέπει να έχουμε έτοιμα και τα πρακτικά και το κείμενο ε, και να τα στείλουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια ούτως ώστε να ξέρουν τι συζητήθηκε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλα αυτά θα κάνουμε και να προετοιμάσουμε τις εργασίες του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου. Την Πέμπτη, μην ξεχνάτε ότι θα συζητήσουμε θέματα καταναλωτών, ε, πολιτικής των καταναλωτών, εφαρμογής των νομοθετημάτων ε, με τα εθνικά κοινοβούλια. Επομένως, είναι σημαντικό να προωθήσουμε τις εργασίες μας σε αυτόν τον τομέα μπορώ να σας δώσω τον λόγο για κάποιες σύντομες παρεμβάσεις. Δεν θα ήθελα σήμερα να γίνει μια μεγάλη συζήτηση, γιατί πολλά από τα θέματα έχουμε συζητήσει ούτως ή άλλως και στη διαβούλευση και στην ακρόαση. Και σήμερα είναι η τελική σύνοδος, της, ε, η τελική συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα τώρα οι πολιτικές ομάδες από εδώ και πέρα να αποφασίσουν τι κείμενο θα πάει στην ε, Ολομέλεια. Δύο ομιλητές, ο κ. Χάρμπορ και η κυρία Γουόλης μόνο. Ε, πολύ ωραία τα συνοψίσατε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θα ήθελα απλώς να ενδυναμώσω αυτά που είπατε και να υπογραμμίσω αυτά που είπατε σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Φερχόγγεν πριν από λίγο. Ξοδέψαμε αρκετό χρόνο να μελετήσουμε την μελέτη επιπτώσεων και τους στρατηγικού, αν θέλετε, προβληματισμούς τη επιτροπή που στηρίζουν την πρόταση. Νομίζω ότι αυτά μας βοηθούν για να έχουμε και εμείς μια στρατηγική προσέγγιση σε αυτή την ε, πρόταση. Όλα αυτά, αυτό, το έργο, ας πούμε, θα το παραδώσουμε στους διαδόχους μας. Επίσης παρατήρησα ότι τονίσατε ότι είναι η τελευταία συνεδρίαση και ότι αύριο το βράδυ θα πιούμε κάποια αποχαιρετιστήρια ποτά, ας πούμε. Έχουμε και την 27η Απριλίου είχαμε τουλάχιστον μια συνεδρία στις 27 Απριλίου. Αλλά μάλλον δεν νομίζω ότι ισχύει αυτή η ημερομηνία τελικά. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί τελικά στην Ολομέλεια του Απριλίου. Σε ποια Ολομέλεια ακριβώς, για πέστε μας. Θα, θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα και τι πρέπει να περιμένουμε, πώς να προετοιμαστούμε, διότι καλό θα ήταν πριν φτάσουμε στην προφορική ερώτηση να συζητήσουμε το θέμα και στις πολιτικές ομάδες. Θα έχουμε χρόνο. Δεν θα περάσει το θέμα στην ε, Ολομέλεια του Απριλίου. Ούτως ή άλλως ε, οι πολιτικές ομάδες αποφάσισαν να μην ε, υποβληθούν προφορικές ερωτήσεις στην Ολομέλεια του Απριλίου. Θα πάει το θέμα αυτό στην τελική Ολομέλεια αυτού του Κοινοβουλίου και επομένω, θα έχουν χρόνο και οι πολιτικέ ομάδε να συζητήσουν αυτό το θέμα. Στις 27 Απριλίου. Αυτό το θέμα, ε, αυτή την ε, ημερομηνία την έχουμε κρατήσει ακόμα ανοιχτή. Είναι μια απόφαση που πήραν οι συντονιστέ. Θα ξαναδούμε αν χρειάζεται πραγματικά να γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής. Σας είπα τώρα ότι η προφορική ερώτηση είναι θέμα των πολιτικών ομάδων και όχι της ε, Επιτροπής γιατί ουσιαστικά δεν υπογράφουμε μια έκθεση που θα υποβληθεί στην Ολομέλεια, αλλά μόνο μια προφορική ερώτηση. Επομένως, θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να αποφασίσουν για το περιεχόμενο της ε, προφορικής ερώτησης. Δεν χρειάζεται λοιπόν ε, να ξανασυνεδριάσουμε ως Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά έχουμε έτσι ανοιχτή την ημερομηνία της 27ης Απριλίου. Εμείς θα αποφασίσουμε. Δεν έχουμε ακυρώσει ακόμα αυτή την ημερομηνία. Κύριε Γουόλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που την περασμένη εβδομάδα απουσίαζα από το Στρασβούργο. Φυσικά ήταν το έγγραφο εργασία και μετά από τις σημερινές σας εξηγήσεις καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εμπεριστατωμένο. Ένα σημείο έχω να υπογραμμίσω. Και έχει να κάνει και με τη δουλειά που κάνω στην Επιτροπή μια βασική έννοια, ότι αν υιοθετήσουμε αυτή την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τότε, όπως είπαν και κάποιοι ομιλητές στην ακρόαση, τότε αποσπούμε το δίκαιο για τους καταναλωτές από το γενικό εταιρικό δίκαιο. Αν κάνουμε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να την κάνουμε με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και θα πρέπει να γνωρίζουμε και τις επιπτώσεις. Στο διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια την Πέμπτη θα πρέπει να το συζητήσουμε γιατί θα τους ενδιαφέρει τα μάλλα αυτό το θέμα. Επομένως κάπως πρέπει να μπει αυτό το θέμα στο έγγραφο εργασίας, να το στριμώξουμε. Είναι μια πολύ σημαντική έννοια. Είναι ουσιαστικά ένα σημείο αφετηρίας θα έλεγα για όλη την οδηγία. Εσείς είδατε μόνο το προσχέδιο του κειμένου. Ε, γι' αυτό δεν υπάρχει και μπροστά σας ε, σήμερα. Είχαμε πει ότι, ότι όποιος συνάδελφος θέλει να κάνει τροπολογίες θα έπρεπε να τις είχε στείλει μέχρι την περασμένη Παρασκευή για να τις συμπεριλάβουμε. Εμείς λέμε ότι αν υιοθετήσουμε αυτή την άγουσα φυσικά θα υπάρχουν επιπτώσεις. Είναι μια πολιτική απόφαση όχι ακόμα, εμεί δεν την έχουμε πάρει. Κάποια στιγμή θα λυθεί όμω αυτή η πολιτική απόφαση. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα την πάρουμε αυτή την πολιτική απόφαση ή θα περιμένουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε πολύ. αν θα πρέπει να περιμένουμε δηλαδή το κοινό πλαίσιο αναφορά. Αν πρέπει να το περιμένουμε, μπορεί να χρειαστούν και 10 ή 20 χρόνια για να συμφωνήσουν κάποια κράτη-μέλη. Σα είπα ότι αυτό το κείμενο δεν είναι μια πολιτική απόφαση, δεν μα δεσμεύει στο μέλλον. Ο κ. Φαμπ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς όμως ο κύριος Φαμπ. Ναι, τώρα εντάξει. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο συντάχθηκε το έγγραφο με μεγάλο πνεύμα συμβιβαστικό και πριν τις ευρωεκλογέ είναι καλό να διατηρήσουμε τη διαδικασία σε αυτό το θέμα, να αναγνωρίσουμε από κοινού ότι έχει μεγάλες αδυναμίες, χωρίς όμως να απεμπολίσουμε την πεποίθησή μας ε, που λέει ότι χρειαζόμαστε στο αστικό δίκαιο κάποια στιγμή μια νέα ρύθμιση για τους καταναλωτές. Νομίζω ότι είναι καλή βάση αυτή και στην επόμενη θητεία θα έχουμε ε, καλή ακριβώ βάση και θεμέλια για να οικοδομήσουμε εκεί τη συνεργασία μας. Ωραία. Αν είναι αυτά όλα τα σχόλια, να θεωρήσουμε ότι λίγη εδώ αυτή η συζήτηση. Έχουμε όλα τα σχόλια, όλες τις θέσεις των συναδέλφων θα ολοκληρώσω το προσχέδιο αυτή την εβδομάδα και αμέσως περίπου θα έχουμε ε, γαλλικά και γερμανικά. Κάποια στιγμή θα έρθει σε όλες τις γλώσσες μέχρι την Ολομέλεια, στη δεύτερη του Μαΐου και στο μεταξύ θα χρησιμοποιήσουμε το έγγραφο για να συντάξουμε την προφορική ερώτηση. Δεν θα σας εκπλήξει τίποτα γιατί απορρέει από τα όσα γράφει το έγγραφο εργασίας. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τις τοποθετήσεις σας και προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι μια παρουσίαση της Χότρεκ για την πυρασφάλεια στα ξενοδοχεία. Θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους πώς φτάσαμε ως εδώ. Η κυρία Μαργαρίτσα Χάρου που είναι η αρμόδια θα κάνει την παρουσίαση. Ξέρετε ότι πριν από καιρό μας ζητήθηκε μάλλον ζητήσαμε εμείς να κάνουμε κάποια δουλειά και για το μονοξίδιο του άνθρακα και για τις δοκιμές. Το κάναμε αυτό γιατί δεν έχουμε νομοθεσία, ε, ούτε νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά μια σύσταση του Συμβουλίου του 1986 για την πυρασφάλεια στα ξενοδοχεία και πολλές οργανώσεις και καταναλωτών απευθύνθηκαν σε μας και διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν εφαρμόζεται, λέει, από τα κράτη-μέλη από το 86 αυτή η σύσταση και θέλανε λίγο περισσότερη δουλειά να κινηθούν τα πράγματα. Και πιστεύουμε εδώ στην Επιτροπή μας ότι χρειάζεται να γίνει αυτό, γιατί όλοι ζητούμε από τους καταναλωτές να ε, πηγαίνουν σε διάφορα τέτοια ξενοδοχεία, θέρετρα, διασυνοριακή υπαροχή υπηρεσιών και αυτό που θα ε, περίμενε κανείς το ελάχιστο είναι να υπάρχουν ασφαλείς προδιαγραφές. Υπήρξε ένα εργαστήριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για, ε, ε, μάλλον που ανέθεσε μια μελέτη για να δούμε τι γίνεται. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμφωνήσατε και ο κλάδος να το προωθήσει ως κώδικα συμπεριφοράς ή χάρτα ασφάλειας και χαιρόμαστε που ήρθαν σήμερα εδώ από τη Χότρεκ να μας ενημερώσουν για το χρονοδιάγραμμά του τι προτάσει του, και χωρί άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στην κυρία Σικάρη. Σα σωστά λέω το όνομά σα. Okay. Corporate... Και ο κύριο Paul Μόξ που είναι αντιπρόεδρος ε, στον Όμιλο Ρεζιντόρ και ο κύριος Αλέξης Βαράφκα είναι πολιτικό σύμβουλος της Χότρακ. Έχουμε πολλούς εκπροσώπους να μας βοηθήσουν εδώ σήμερα. Παρακαλώ. Καλώς ορίστε στην Επιτροπή μας και ελάτε σας παρακαλώ λάβετε το λόγο. Of the Parliament. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, ε, σας ευχαριστώ μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο μας στην Επιτροπή σας. Εκπροσωπούμε την ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξενοδοχείων, Καφέ και Εστιατορίων όπως σας είπε και η κυρία Πρόεδρος, ο κύριος Πολ Μόξνες εκπροσωπεί το Group Residor, δηλαδή εκπροσωπούμε και εθνικές ε, ενώσεις και μεγάλες αλυσίδες. Η Χοτρέκ ε, είναι μια συνομοσπονδία 40 εθνικών ομοσπονδιών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του κλάδου σε 25 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος πάντων δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω με αυτά, θα περάσω αμέσως το κύριο μέρος του έργου μας. Εμείς είδαμε τι γίνεται με το τι υπάρχει στον τομέα. Είχαμε μία σύσταση 1986, την οποία ακολούθησαν πάρα πολλοί κανόνες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ε, επί χρόνια συζητούσαμε την δυνατότητα αναθεώρησης της σύστασης του 86, αλλά χωρίς επιτυχία. Παρόλα αυτά υπάρχει αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν να επανεξεταστεί το ζήτημα. Οπότε η συνομοσπονδία μας δέχτηκε να εξετάσει το ζήτημα και να ξεκινήσει ένα έργο με στόχο να βελτιωθεί η πυρασφάλεια των ξενοδοχείων στην Ευρώπη και για να γίνει αυτό χωρίς περισσότερους κανονισμούς και να γίνει αυτό και προς ε, το συμφέρον μικρών και μεγάλων εταιριών, μεμονωμένων και αλυσίδων, υπαρχόντων και καινούριων και με στόχο να καλύψει όλες τις ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό στενή συνεργασία με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Οπότε καταλήξαμε σε ένα ευγερσιακό σχέδιο που ενέκριναν όλες οι εθνικές μας ομοσπονδίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπευλήθη άτυπα στο τελευταίο εργαστήριο της Επιτροπής σας, όπου αναλύθηκε η μελέτη ασφαλείας και χαιρόμαστε που σήμερα είμαστε εδώ για να σας μιλήσουμε πιο επίσημα, αν θέλετε, για το έργο μας αυτό. Ποια είναι τα παραδοτέα εδώ πέρα. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα μία χάρτα που θα πρέπει να υπογράψουν όλες οι εθνικές ομοσπονδίες, μέλη μας και θα αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για καλύτερη πυρασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χάρτα η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σύγχρονη μεθοδολογία δομημένη γύρω από τρία γράμματα. Τα MBS στα αγγλικά, δηλαδή διαχείριση, management ε, B αντιστοιχεί στο building features τα χαρακτηριστικά της οικοδόμησης και F για fire safety τα συστήματα πυρασφάλειας. Οπότε αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε το έργο εντός της ομάδας εργασίας της Συνομοσπονδίας μας και θα επανέλθουμε με τη θέση αυτής της ομάδας εργασίας τα ευρήματα της οποίας θα πρέπει να παρουσιαστούν και να ενισχυθούν από μια συμβουλευτική επιτροπή ενδιαφερομένων μερών και θα σας εξηγήσω ποιοι συμμετέχουν σε αυτή και μετά θα έχουμε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσής μας, δηλαδή όλων των Εθνικών νομοσπονδιών που είναι μέλη μας, γιατί σημαντικό είναι να μην συμφωνήσουμε μόνο εμείς εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά η χάρτα αυτή να εφαρμοστεί ε, σε όλα τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι πρώτης, ε, πρώτη πρώτου του 2010. Τώρα, για την ομάδα εργασία είναι μια ομάδα εργασία της ομοσπονδία μας. Μέλη και πρόεδρος είναι όλοι μέλη των Εθνικών Ομοσπονδιών που έχουν σοβαρή πείρα στον τομέα της πυρασφάλεια. Έχουμε λοιπόν και εκπροσώπους από πολλές χώρες και εκπροσώπους αλυσίδων. Είναι εδώ ο κύριος Πολ Μόξνες που αντιπροσωπεύει όπως σας είπα δίκτυο και από μεμονωμένα ξενοδοχεία. Μας ε, βοήθησε λοιπόν ο Πάτρικ Κάρεϊ, ο οποίος είναι πεπειραμένος σύμβουλος πυρασφάλειας ε, στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο και ένας ανεξάρτητος εκπρόσωπος, ο κύριος Ντίτερ Νίσλερ, που είναι στέλεχος της πυροσβεστικής. Οπότε, επίσης ενεπλάξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ευρωβουλευτές, οι καταναλωτές, η Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιριών, Tour Operators, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πυρασφαλείας, που αποτελείται από δημόσιες αρχές, η Spinklers, η Ένωση Κατασκευαστών Πυροσβεστικών Ειδών και η Ευρωπαϊκή Πυροσβεστική Ακαδημία. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτή τη χάρτα ακόμη είναι στο στάδιο τη συζήτηση. Σκοπεύουμε να υπογραφεί από όλε τι εθνικές μας ομοσπονδίε. Πρέπει να είναι απλή και σύντομη και να επικεντρώνεται σε αυτό το οποίο εμεί θεωρούμε πυλώνε τη ορθής διαχείρισης ε, των ξενοδοχείων. αν θα είναι 7 ή 8 οι πυλώνε, θα το δούμε. Μέχρι στιγμής έχουμε καταλήξει 7, σε 7 πυλώνες, δηλαδή να υπάρχει υπεύθυνο πυρασφάλειας, να υπάρχει ένα αρχείο πυρός, να υπάρχει ένα σχέδιο ανταπόκρισης, εκπαίδευση του προσωπικού, να υπάρχει άσκηση πυρασφάλειας τουλάχιστον μια φορά το έτος, συντήρηση και επιθεωρήση του εξοπλισμού και της αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς. Σε τι θα δεσμευτούν τώρα οι ε, υπογράφοντες. Θα ενθαρρύνουν τα μέλη τους τα ξενοδοχεία δηλαδή μεμονωμένα οι αλυσίδες που συμμετέχουν να δεσμευτούν σε αυτές τις 7 αρχές και η Εθνική Ένωση μετά θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα στήσει μία βάση δεδομένων θα προωθήσουν τη χάρτα και τη νέα μεθοδολογία αυτή στις ε, ε, κρατικές αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είτε αυτές ε, ασχολούνται από την πλευρά της ε, νομοθεσίας είτε από την πλευρά της επιθεώρησης και βεβαίως ε, θα ε, αναφερθούμε μετά. Θα δώσουμε αναφορά και στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Επίσης, η μεθοδολογία αυτή η οποία ακόμα είναι υποσυζήτηση θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο φιλικό προς την διαχείριση του ξενοδοχείου. Ως βάση θα έχουμε διάφορα έντυπα που έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή στις εθνικές μας ομοσπονδίες, είτε εντό κάποιων ομίλων όπως η Ρεζάιντορ. Επίσης γίνεται και υπό την καθοδήγηση του κυρίου Πάτρικ Κάρι και όταν προχωρήσει αρκετά θα προταθεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή των Διαφερόμενων για τα σχόλιά τους. Λίγα λόγια ακόμα για τη μεθοδολογία μας αυτή του MBS όπως σας είπα αλλά θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στο M αυτής τριάδας στην διαχείριση δηλαδή γιατί είναι κρίσιμη και εκεί πέρα θα αναπτύξουμε τις 7 ή 8 αναλόγως αρχές της ορθής διαχείρισης ξενοδοχείων που θα αναπτυχθούν στη χάρτα μας γιατί θεωρούμε βεβαίω πως η διαχείριση είναι η βασική πτυχή της αύξησης πυρασφαλείας στην Ευρώπη. Εδώ πέρα βλέπετε το χρονοδιάγραμμα. Όπως σας είπα, είμαστε στα πλαίσια της ομάδας εργασίας αυτή τη στιγμή. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα συνεδριάσει αρχές Ιουνίου και το Σεπτέμβριο μετά ξανά. Και ελπίζουμε να εγκριθεί το έργο συνολικά το φθινόπωρο, μετά να το παρουσιάσουμε σε Κοινοβούλιο και Κομισιόν πριν το τέλος του έτους και να ξεκινήσει πια εφαρμογή αρχές του 2010. Εάν έχετε προτάσεις, σχόλια, Ευχαριστώ να τα ακούσουμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Πολ Μόξνες, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός εμπειρογνώμονας εγώ έκανα τα εύκολα, ο κύριος Μόξτεν λοιπόν θα κάνει τα δύσκολα. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ χρήσιμα αυτά και να έχουμε και μια προοπτική χρονική έτσι για τα όσα μας λέτε. Δεν ξέρω αν έχουν ερωτήσεις οι συνάδελφοι για την παρουσίαση αυτή. Έχετε ερωτήσεις? Εγώ σημείωσα ότι όπως ζητήσαμε Καλύψατε τα ιστορικά κτίρια, τα υπάρχοντα φυστάμενα και τα επόμενα. Ερωτήσεις δεν έχετε, συνάδελφοι. Ε, γιατί έχω εγώ τότε, έχω δύο ειδικέ ερωτήσεις. Αυτή η χάρτα που προωθείτε και θα προσυπογράψουν διάφορα μέρη. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να δω πώς θα λειτουργήσει αυτή. Τι σημαίνει για μένα αυτός κατά ανανότρια. Αν είναι δεσμευτικό ο χάρτη αυτός, εγώ θα έχω εγγυήσεις ότι θα υπάρχουν υψηλά πρότυπα πυρασφάλεια στα ξενοδοχεία. Εγώ που είμαι καταναλώτρια. Ωραία, θα φτιάξετε ένα χάρτη, μια χάρτα, πώς τη λένε. Εμένα τι θα μου ε, ε, αποφέρει αυτό ως καταναλώτρια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεύτερον, θα θυμάστε ότι ένα από τα ζήματα που ετέθησαν και δεν αναφέρονται στην παρουσίασή σας ήταν ότι ανησυχούσαν κάποια συνάδελφοι για το μονοξίδιο του άνθρακος που είχαμε ε, ε, δηλητηρίασεις. Ε, ξέρω δεν το γράφει αυτό ε, η μελέτη σας. Θα μπορούσε όμως να καλυφθεί γιατί είναι θέμα ασφάλειας, έτσι, πέρα από την πύρα ασφάλεια. Κύριε Χάρμπορ, δεν έχετε ερωτήσει για την πρόταση. Ε, όχι, δεν έχω. Καλά. Μήπως να απαντούσατε τότε σε μερικές από τις δικές μου ερωτήσεις. Well, thank you for... Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω. Στην ομάδα μας είχαμε τον εξής λόγο για να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια. Επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε συνειδητοποιήσει ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια στα ξενοδοχεία μας, εξαρτώμεθα από την προσπάθεια που κάνει κάθε υπάλληλο ξενοδοχείου σε κάθε επίπεδο. Όπου και αν βρίσκονται τα ξενοδοχεία μας. Όμως τα ξενοδοχεία που έχουμε είναι τόσο διαφορετικά σε ό,τι αφορά τη δομή τους, εσωτερική οργάνωση, νομικό πλαίσιο, την ηλικία τους. Δεν μπορούμε να κάθομαστε στα γραφεία μας και να εκπονήσουμε ένα εγχειρίδιο για όλα τα ξενοδοχεία. Γι' αυτό λοιπόν μια χάρτα η οποία θα μας βοηθούσε να οργανώσουμε τις προσπάθειές μας, θα μας βοηθούσε πολύ περισσότερο γιατί θα γινόταν στα ξενοδοχεία. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Και αυτό θα είναι επωφελές και για τους καταναλωτές και για τους υπαλλήλους, που και αυτοί κινδυνεύουν στα ξενοδοχεία λόγω πυρκαγιάς. Όταν Καταρτίζουμε τους υπαλλήλους μας, τους ρωτάμε να μας πούν γιατί έχουμε ανιχνευτές στα ξενοδοχεία μας. Και αυτοί πάντα απαντάνε ότι τους έχουμε για την ασφάλεια των ανθρώπων που διαμένουν στα ξενοδοχεία. Αλλά οι πελάτες μένουν ένα-δύο βράδια. Οι υπάλληλοι δουλεύουν μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Επομένως, ε, αν το δείτε το θέμα αυτό από στατιστικής ε, σκοπιάς, το κινδυνεύουν οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου παρά οι πελάτες. Επομένως, αν οι αφυπνιστούν οι υπαλλήλοι μας για τα θέματα ασφάλειας του ξενοδοχείου, αν ε, ελέγξουν τα θέματα ασφάλειας και αν συνειδητοποιήσουν το κάνουμε για τη δική τους ασφάλεια, νομίζω ότι προχωρούμε πολύ περισσότερο από ότι αν επενδύσουμε πάρα πολύ σε τεχνικό εξοπλισμό. Και το όφελος για τους καταναλωτές θα προέλθει από την μεγαλύτερη συνείδηση που υπάρχει στους υπαλλήλους μας και με αυτόν τον τρόπο διαχειριζόμαστε τα θέματα ασφάλειας με καλύτερο τρόπο και στα ξενοδοχεία. Ελπίζω να σας απάντησα. Φυσικά θέλουμε να σε ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Χαιρόμαστε που εκπονείται αυτή τη χάρτα. Το θέμα είναι που μπαίνει εδώ ο καταναλωτή. Γιατί φυσικά δεν είναι θέμα μόνο καταναλωτών εδώ, είναι και θέμα ε, εργαζομένων. Αν εγώ κλείσω μία νύχτα σε ένα ξενοδοχείο, θα ήθελα να ξέρω ε, αν ε, το ξενοδοχείο αυτό έχει προσυπογράψει αυτή τη χάρτα. Ε, επομένως, να είμαι σίγουρη ότι κρατάει ψηλά το επίπεδο της πυρασφάλειας να υπάρχει κάποιος υπεύθυνο για την πυρασφάλεια, κάποιος στον οποίο να μπορώ να απευθυνθώ, όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρεται. Να έχουμε λοιπόν αυτή την εγγύηση ασφάλειας ως καταναλωτές. Και κάτι άλλο, μια τελευταία ερώτηση. Το θέμα της δηλητηρίασης από το μονοξίδιο του άνθρακα είναι θέμα ή δεν είναι. Θα πρέπει να μπει σε αυτό το πακέτο ασφάλειας. Ε, εσείς αποφασίσατε να μην το βάλετε. Ε, και το, το θέτω αυτό το ερώτημα γιατί το ενδιαφέρει και διάφορου συναδέλφου. Το έθεσαν και διάφοροι συναδέλφοι. Ζητώ συγγνώμη που δεν σα απάντησα αυτό το δεύτερο ερώτημα για το μονοξίδιο του άνθρακα. Στα έγγραφα που εκπονούμε, έχουμε ετοιμάσει και ένα τμήμα για το μονοξίδιο του άνθρακα. Δεν το τονίσαμε στη σημερινή παρουσίαση, αλλά το έχουμε λάβει υπόψη μας. Και οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες, όπως αυτή που εκπροσωπώ, ε, έχουν λάβει υπόψη τους το μονοξίδιο του άνθρακα ως τμήμα του προγράμματος ασφάλειας του ξενοδοχείου τους. Το πώς αναγνωρίζεται αυτό τώρα στην κράτηση, μπορούμε να κάνουμε την κράτηση με διαφορετικούς τρόπους, αλλά όλα τα ξενοδοχεία που είναι μέλη μιας διεθνούς οργάνωσης που έχει προσυπογράψει αυτή τη χάρτα, φυσικά, επειδή είναι μέλη της χάρτας, δεν έχουμε μπει σε λεπτομέρειες ακόμα, αλλά θα υπάρχει μια αναφορά στα έγγραφα κράτησης του ξενοδοχείου και νομίζω ότι είναι ένα καλό διαφημιστικό κόλπο και ένα καλό στοιχείο μάρκετινγκ για το ξενοδοχείο. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο, λέει η Πρόεδρος. Γιατί το έχουμε συζητήσει και με την Κομισιόν αυτό το θέμα. Το έχουμε θέσει και στην Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτά που ακούσαμε σήμερα όντως έχουν συζητηθεί και στην Κομισιόν και με την Κομισιόν και με αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και ήμασταν όχι μόνο παρόντες, αλλά είχαν οργανώσει την συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Ενδιαφερομένων και την, ε, τελευταία συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής ε, εκπροσωπήθηκε και η κοινοβουλευτική σας επιτροπή. Νομίζω ότι μπορείτε να εκπροσωπηθείτε και σε επόμενες συνεδριάσεις που θα γίνουν. Ως προς το συγκεκριμένο σας ερώτημα, πώς θα καταλάβω εγώ ως καταναλωτής ότι τα πράγματα είναι εντάξει για μένα, ότι είμαι ασφαλής. Το είχα θέσει αυτό το ερώτημα στην πρώτη συνεδρίαση των ενδιαφερομένων. Η απάντηση που έλαβα από τη ήταν καθησυχαστική σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση. Τι διατάξεις παρακολούθησης θα υπάρχουν για όλους όσους προσυπογράφουν τη χάρτα. Φυσικά ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες πάντα. Θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται αυτή η παρακολούθηση, πώς εξελίσσεται σύντο χρόνο. Αλλά υπάρχουν αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία νομίζω Νομίζω ότι τα ξενοδοχεία πραγματικά αναλαμβάνουν αυτές τις δεσμεύσεις και τις αναλαμβάνουν στα σοβαρά. Στις πρώτες συνεδριάσεις ε, της... που οργανώσαμε ήταν ε, εκπρόσωπος ε, της οργάνωσης των Ευρωπαίων Tour Operator είπαν ότι θα καταστήσουμε υποχρεωτική την υπογραφή της χάρτας προκειμένου να δεχτούμε τα ξενοδοχεία αυτά να συμμετέχουν στα προγράμματα των δικών μας tour operator. Αυτό ήταν πολύ καθυσυχαστικό. Και νομίζω ότι αυτό θέλει και ο Επιτροπός μου και η Επιτροπή σας. Πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, και ως καταναλωτής που τα παρακολούθησα πάρα πολύ προσεκτικά αυτό το το θέμα, θα θέλαμε πραγματικά να υπάρχει προϋπόθεση υπογραφής της χάρτας. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει αυτός ο εθελοντικός κώδικας, αυτή η εθελοντική ρύθμιση, καλό είναι ε, να μιλήσουμε για το επίπεδο των προτύπων που θα θέλαμε να υπάρχει. Και να προωθηθεί αυτή η χάρτα ούτως ώστε εγώ ως καταναλωτής να ξέρω αν το τάδε ξενοδοχείο ε, έχει προσυπογράψει τη χάρτα ή όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ξέρετε ότι οι οργανώσεις των ταξιδιωτών θέλουν νομοθεσία σχετικά. Έχουμε τη σύσταση του 1986. Αν μακροπρόθεσμα δούμε ότι αυτή η προσπάθεια δεν γενικεύεται, νομίζω θα υπάρχουν ε, στεναρά επιχειρήματα από τις οργανώσεις ταξιδιωτών ε, για να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό δίκαιο. Μια πρόταση δηλαδή νομοθετικού χαρακτήρα. Σήμερα λοιπόν σας ευχαριστούμε που κινείστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, σας υποστηρίζουμε, θα συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε και θα σας ε, βοηθήσουμε να προωθήσετε αυτό το εγχείρημα, ούτω ώστε να ανεβούν τα πρότυπα και η προστασία των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα περιμένουμε και τα... τις επόμενες συναντήσεις ενημέρωσης και θα θέλαμε να, συνεδρι... να συμμετάσχουμε κι εμείς στη συνεδρίαση των ε, stakeholders φυσικά. Ο κ. Χάρμπορ. Ένα, μία έκθεση για τις σημαντικές διαπραγματεύσεις στις οποίες ε, συμμετείχατε ε, εκ μέρους της Επιτροπής για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις υπηρεσίες για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας ε, σας δίνω το λόγο για να μας μιλήσετε για τις τροπολογίες. Ε, κάποιοι από τους γεώδεις ηγητές είναι εδώ, δεν είναι όλοι. Ξέρω ότι συνομιλούσατε μαζί του σε τακτή, βάση, επομένως <laughs> δεν με ανησυχεί αυτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε κάποιες συμβαστικέ τροπολογίες, τι διαπραγματευτήκαμε αυτές και ελπίζω να σας έχουν μοιραστεί ή θα σα μοιραστούν. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν τις έχετε έφτασε εδώ ο Πίτερ με τις τροπολογίες. Τις έχουμε λοιπόν αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Λοιπόν, ας τις διατρέξουμε. Θα ήθελα παρακαλώ να μοιραστούν και τα κείμενα στους βουλευτές. θα μιλήσω για τη διαδικασία, για το που βρισκόμαστε πριν τις τροπολογίες. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες εισηγητές και όλο το προσωπικό που μας πλαισίωσε για αυτή την πρόταση, γιατί δουλεύουμε για αυτή την πρόταση αρκετούς μήνες τώρα, ε, μετά τη συμφωνία της κοινή θέση. Και είχαμε ξεκινήσει μάλιστα τη δουλειά και πριν την κοινή θέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πακέτο των τηλεπικοινωνιών και τη θέση μας. Ε, έχω συνεργαστεί με τους ε, εισηγητές ε, των άλλων επιτροπών πολύ στενά και με το Συμβούλιο για να συμφωνήσουμε σε δεύτερη ανάγνωση, βασιζόμενη πάντα στην κοινή θέση. είχαμε εμπλακεί σε δύσκολες, μακρές, χρονοβόρες διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η θέση του Κοινοβουλίου ε, απεικονίζεται καλύτερα στην κοινή θέση. Τώρα, η πολιτική προτεραιότητα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, εστίαζε καταρχάς στις οικονομικές ε, ρυθμίσεις και κανόνες και στο, στην ύπαρξη ενός νέου ρυθμιστικού σώματος το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν φτάσει ουσιαστικά συμφωνία για αυτό το θέμα. Εγώ είχα εμπλακεί σε αυτέ τι διαπραγματεύσει για κάποια θέματα που ενδιαφέρουν κυρίω αυτή την Επιτροπή. Δεν μπορώ να ήξερα τι λεπτομέρειε, φυσικά δεν έχουμε πιο χρόνο. Και ε, μάλλον θα έχουμε τον τελικό τριμερή διάλογο σήμερα το βράδυ. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ιδιωτική σφαίρα, ε, στη συζήτηση του Συμβουλίου δεν είχαν την πρωτοκαθεδρία, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες ε, είχαμε έντονες ε, συζητήσεις για τις προτάσεις για τα δικαιώματα των χρηστών. Και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει θετικά βήματα υπέρ των καταναλωτών σε σχέση με την πρώτη ανάγνωση. Θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για την επικοδομητική προσέγγιση που είχε στις διαπραγματεύσεις. Ο λόγος που δεν προχωρήσαμε περισσότερο είναι ότι όχι δεν θέλουμε να φτάσουμε σε συμφωνία, αλλά δεν είχαμε αρκετό χρόνο μαζί, γιατί είχαμε τρία, τρεις φακέλους που συζητούσαμε παράλληλα. Την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε πολύ από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Η θέση λοιπόν που φτάσαμε ποια είναι. Είναι να σας συστήσω την υιοθέτηση διαφόρων συμβαστικών τροπολογιών που έχουν προσυπογραφεί από όλε τι πολιτικές ομάδες που έχουν εμπλακεί άμεσα, με την εξαίρεση των πρασίνων που έχουν κάποιε επιφυλάξει για τις λεπτομέρειε. Και νομίζω ότι εν γέννη παρόλα αυτά και οι πράσινοι ε, είναι ικανοποιημένοι, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να τις υπεψηφίσουμε αύριο, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να υποβληθούν όλες οι τροπολογίες που είχαν υποβάλει στην αρχικά για δεύτερη ανάγνωση. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, επειδή δεν έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τις τροπολογίες πρώτης ανάγνωσης και υπάρχουν και κάποιοι τομείς όπως ε, την ε, φορητότητα του αριθμού ή τη μεταφορά του αριθμού όταν οι καταναλωτές αλλάζουν πάροχο. Εκεί δεν έχουμε συμφωνήσει, αλλάζουμε το κείμενο, ήταν πολύ δύσκολο θέμα. Ε, έχουμε τροπολογίες λοιπόν. Υπάρχουν δύο κρίσιμες ε, περιοχές για την οδηγία ε, για την ηλεκτρονική ιδιωτική σφαίρα που αφορά την πρόταση για την κοινοποίηση παραβίας των δεδομένων και την διατάξη για το opt-in σε σχέση με το opt-out για να επιτρέψουμε μια εταιρεία να έχει πρόσβαση ε, σε δεδομένα στον υπολογιστή σας, ε, νομίζω ότι υπάρχει μια διατύπωση που θα μας επιτρέψει να διατηρηθεί το opt-in. Θέλουμε να συμφωνήσουμε και για τα δύο αυτά θέματα, αλλά είναι πολύ ευαίσθητα νομικά θέματα εν γέννη. Συνολικά πάντως, ε, σε σχέση με βασικά θέματα προστασίας των καταναλωτών, έχουμε σημειώσει ουσιαστική πρόοδο και τώρα θα ήθελα να περάσω στις συμβαστικές τροπολογίες για να σας πω τι εμπεριέχουν. Θα ήθελα να σας ε, τις σχολιάσω και συνεχεία θα ακούσω τις παρατηρήσεις σας ε, εν ώψη της αυριανής ψηφοφορίας. Λοιπόν, έχουμε, έχουμε τώρα το πακέτο των συμβαστικών λύσεων στα αγγλικά. Πρώτα απ' όλα στη συμβαστική λύση 1 συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο σε μια νέα τροπολογία που θα δώσει περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για να μπορούν να εισάγουν ε, σε απαιτήσει καθολικής ε, παροχής υπηρεσία που τώρα έχουν μια νέα προσέγγιση ευρυζωνικότητας αντί για την προσέγγιση από το 2001 που ήταν, ε, δεν ήταν ευρυζωνική. Οπότε έχουμε μια αλλαγή στο, στο άρθρο αλλά υπάρχει απαραίτητη ευελιξία. Επίσης θέλουμε να πιέσουμε την Κομισιόν έτσι ώστε η αναθεώρηση αυτών των υποχρεώσεων καθολικής παροχής υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί γρήγορα για να μην φτάσουμε στον Ιανουάριο του 2010. Εναλλακτικά η Κομισιόν μπορεί να κάνει μια ξεχωριστή δήλωση για αυτό το θέμα, αλλά εμείς νομίζουμε πως καλό θα ήταν να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο αύριο για να δείξουμε την αποφασιστικότητα της Επιτροπής μας για την ε, προθεσμία. Τώρα υπάρχουν κάποιες διατάξεις ε, με την συμβαστική τροπολογία 2 για τον ε, εξοπλισμό στο τέρμιναλ και δεν ξέρουμε αν είναι σωστό το να φτάνουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας. Θα επανέλθω σε λίγο με τα δικαιώματα των αναπήρων χρηστών που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας. Τώρα να περάσω στη συμβαστική τροπολογία 3. Συμφωνήσαμε πως για να μην καταστεί παροχημένη στο μέλλον η οδηγία η φωνητική τηλεφωνία, η δημόσια φωνητική τηλεφωνία θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από τα τηλέφωνα, τα καρτοτηλέφωνα, γιατί θα έπρεπε να είναι, θεωρούμε, κάτι στο μέλλον, το οποίο θα είναι διαφορετικό από τηλεφωνικό θάλαμο. Θα είναι ένα σημείο παροχής πρισιών π.χ. μεσοδιαδικτύου. Οπότε λογικό νομίζω είναι να διευρύνουμε το εύρος αυτής διάταξης με το να συμπεριλάβουμε όχι μόνο, όπως σας είπα, τους τηλεφωνικούς θαλάμους, ως απέτηση των κρατών μελών, αλλά αυτό το οποίο περιγράφουμε ως ε, σημεία πρόσβασης ε, δημόσιας τηλεφωνίας φωνής. Είναι μια λεπτομέρεια αλλά σημαντική νομίζω θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για το ότι αποδέχτηκε την άποψή μας για την πρόσβαση των αναπήρων χρηστών. Η Συμβαστική Τροπολογία 4 περιέχει μια σειρά διατάξεων με τις οποίες έχουμε επαναφέρει τον όρο ισοδύναμο, ενώ το Συμβούλιο ήθελε να φέρει τον όρο συγκρίσιμο αυτό αυτός ο όρο υπάρχει στην οδηγία την ισχύουσα και δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει γιατί είναι και πιο έντονη διατύπωση, αλλά συμφωνήσαμε σε ένα εκτιμώντα το οποίο θα δώσει ένα σαφή ορισμό του τι εννοούμε όταν μιλάμε για ισοδυναμία πρόσβασης των αναπήρων χρηστών. Οπότε το βλέπετε αυτό εκεί. Οπότε έχει επανεισαχθεί εδώ πέρα ο όρος ε, ισοδύναμος ε, εκεί που είχε βάλει το Συμβούλιο συγκρίσιμο. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου πως έχουμε επιτύχει μια ικανοποιητική λύση. Στην ε, δε συμβαστική λύση 5, που είναι αρκετά μακροσκελής, περιέχονται αρκετά πράγματα για τις απαιτήσει πληροφόρησης και διαφάνειας των καταναλωτών στις συμβάσεις και κατά την συνεχή χρήση των ε, υπηρεσιών. Ε, δηλαδή θα πρέπει να πληροφορούνται οι καταναλωτές για την πρόσβαση υπηρεσίες και τυχόν όρους και επίσης ξεκαθαρίσαμε και τη διατύπωση. Οπότε βλέπετε τώρα όσον αφορά τις ε, πληροφορίες πριν την σύμβαση θα γίνει σαφές στους καταναλωτές το εάν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφαλείας και εντοπισμού του χρήστη και επίσης ε, μείωση της πρόσβασης ε, σε κάποιες ε, εφαρμογές ανάλογα με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, κάτι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό στοιχείο γιατί θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια εάν ισχύουν τέτοιοι όροι και επιβάλλονται από κάποιον πάροχο και διαφάνεια δεν σημαίνει πως επιτρέπονται αυτοί οι όροι παρά μόνο εάν ε, ισχύει κάτι τέτοιο με εθνικό δίκαιο ή δίκαιο του ανταγωνισμού αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ε, π.χ. κάποιος να πάρει κάποιο πακέτο κινητής τηλεφωνίας μόνο με φωνητική τηλεφωνία και χωρίς ε, ίντερνετ και πρέπει να περιγραφεί αυτή η δικαιο του αλλα υπαρχουν και αλλες περιπτωσεις πχ καποιος να παρει καποιο πακετο κινητης τηλεφωνιας μονο με φωνητικη τηλεφωνια και χωρις ιντερνετ και πρεπει να περιγραφει αυτη η αυτός ο περιορισμός πρόσβασης και επίσης υπάρξουν διαδικασίες ε, που θα έχει ο πάροχος για να μετρήσει την ε, κίνηση στο δίκτυό του για να μην υπερφορτωθεί το δίκτυο και το τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα της υπηρεσίας και αυτό είναι σημαντικό και πράγματι αρκετοί παροχοί δίνουν τέτοιες πληροφορίες στους καταναλωτές για το πώς μετρούν και διαμορφώνουν την κίνηση για να υπάρχει συνεχής ποιότητα ειδικά όταν μιλάμε για συνδέσεις ευρυζωνικές, που μπορεί να είναι κάποια υπηρεσία τηλεόρασης ή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, όπου απαιτείται π.χ. σύνδεση υψηλής ευκρίνειας, κάτι το οποίο δεν ισχύει π.χ. για τα email αλλά πρέπει ε, ο καταναλωτής να παρατηρεί αλλαγή στην ποιότητα. Και αυτά επιδρούν στην πολύ αυτή ευρεία έννοια της ουδετερότητας του διαδικτύου. Ξέρω πως λαμβάνετε πολλά email από πολλές πλευρές. Εμείς θεωρούμε πως ο συμβασμός μας είναι ξεκάθαρος. Ότι οποιαδήποτε ζητήματα περιορισμού της πρόσβασης ε, και διαδικασίες διαμόρφωσης κίνησης πρέπει να συμμορφώνονται πάντα με, τον κανό, με τους κανονισμούς του δικαίου του ανταγωνισμού περί μη διάκρισης. Πρέπει να δικαιολογούνται και να είναι κυρίως διαφανείς προς τους καταναλωτές και αυτό θεωρούμε ότι είναι ο καταλληλότερος τρόπος. Και σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου εδώ υπάρχει επιλογή παρόχου και πρόσβαση στις υπηρεσίες, θεωρούν πως ε, πράγματι κάτι τέτοιο είναι σωστό. Κάτι το οποίο δεν ισχύει στη ΣΥΠΑ. <coughs> Κάποια δε από τα επιχειρήματα που ακούστηκαν ε, μάλλον αφορούν περισσότερα το περιβάλλον των ΙΠΑ παρά της Ευρώπης. Οπότε εμείς διασφαλίζουμε την ελευθερία πρόσβαση στο ίντερνετ και τα συμφέροντα του Τώρα, δεν θέλω να μπω σε υπόλοιπε λεπτομέρειε για του άλλου όρου που έχουμε, γιατί υπάρχουν και κάποιε άλλε λεπτομερεί αλλαγέ. Βρήκαμε πάντως μια φόρμουλα για σέματα πληροφόρηση. Θα έρθω στη συνέχεια στο άρθρο 21 και σε άλλους τομείς όπου έχουμε λεπτομερείς τροποποίηση συμβάσεων και μια φόρμουλα ε, για τις διαφημίσεις το ε, σημείο ε ή που γίνεται λόγος για ελάχιστη χρήση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται μια αρχική προσφορά για να χρησιμοποιήσετε μερικά λεφτά, λεπτά δωρεάν κτλ. Αυτό όμως να λύγει μετά από λίγο καιρό και δεν είναι σαφές ότι για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα είναι πιο διαφανής. Στο άρθρο 21 για τη διαφάνεια λοιπόν και για τη διάρκεια μιας σύμφασης. Μαζί με το Συμβούλιο βελτιώσαμε σημαντικά και διευκρινίσαμε τις διατυπώσεις για την τιμολόγηση και την ενημέρωση για την ανεξάρτητη ε, εκτίμηση του κόστος ε, των διαφόρων πακέτων χρήσης, ε, υπενθυμίσεις για την τιμολόγηση και εδώ λέμε ότι αν γίνει με οποιαδήποτε αλλαγή στους ε, περιορισμούς της υπηρεσίας ή στις διαδικασίες ή αν αλλάξει δηλαδή τις μεθόδους στην πορεία, τότε είναι υποχρεωμένοι σαφώς να ενημερώνει τους καταναλωτές γι' αυτό. Θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε βάλει μια διάταξη που εμείς ε, ε, σε βάθος ε, τροποποίησαμε. Ότι να μπορούν να ανακοινώνονται διάφορες δημόσιες πληροφορίες και σε συνδρομητές νυν και επομένους. Υπάρχει ένας όρος όμως εδώ. Να γίνεται αυτή η πληροφόρηση μέσω τρόπων ή μέσων που συνήθως χρησιμοποιούν οι εταιρείε δωρεάν ε, και παρέχονται στους δρομητές. Δηλαδή δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να προτείνουν άλλους τρόπους επικοινωνίας πέρα ε, από αυτούς που χρησιμοποιούν για να φτάσουν στους συνδρομητές. Δηλαδή δεν μπορείς να επιβάλλεις επιπλέον κόστος στους καταναλωτές. Επίσης, όλα αυτά τα λέει η αιτιολογική σκέψη 24 για τη σχέση των συμβαλωμένων μερών. Έρχομαι τώρα στη συμβαστική υπαριθμόν 26, που είναι νέα αιτιολογική σκέψη και εκκρεμούν ακόμα κάποιες διαπραγματεύσεις. Και ουσιαστικά εμείς θεωρούμε ότι περιλαμβάνει όλη τη θέση μας για την πρόσβαση επικοινωνίες, για την ποιότητα των υπηρεσιών και τις σημαντικές ε, απαιτήσει να θεωρούνται θεμητές ε, μόνο εφόσον είναι συμβατές οι διάφορες διαδικασίες και να μην υπάρχει προτίμηση σε κάποιες υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος ο πάροχος σε σχέση με κάποιον ανταγωνιστή του. Και έρχομαι τώρα στο άρθρο 22.3 που δεν αλλάξαμε, ένα προαπαιτούμενο εκεί, όπου μπορεί να προτείνεται υποχρέωση παροχής ε, υπηρεσιών. Γιατί μπορεί κάποιος πάροχος υπηρεσίας να κάνει σαμποτάζ, ας πούμε, να, να επιβραδύνει μια υπηρεσία του ανταγωνιστού σε σχέση με τη δική του για να προτιμάει ο καταναλωτής τη δική του. Και εδώ εξετάζουμε αυτά τα μέτρα κατά το διαχρήσεων, λοιπόν. Συμβαστική τυπολογία υπερθμών 7. Έχουμε κάνει σημαντικές αλλαγές εκεί για να βελτιώσουμε, πιστεύουμε, το περιβάλλον της διαφάνειας και του ανταγωνισμού. Στη συμβαστική υπερθμών 8 και αυτό αφορά τη μεταφορά του αριθμού. Χαιρόμαστε μας πάρα πολύ που το Συμβούλιο τα δέχτηκε όλα αυτά που προτείνουμε εδώ για περιορισμό στη διάρκεια της σύμβασης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διετία και επίσης τη δυνατότητα σύμβαση ε, ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Αυτές είναι σημαντικές ε, βελτιώσεις υπέρ των καταναλωτών που δεν περιείχε το αρχικό κείμενο του Συμβουλίου. Πάντως στην παράγραφο 4 για το ε, τη μεταφορά του αριθμού ε, θα χρειαστεί διαπραγμάτευση για μια αιτιολογική σκέψη. Τώρα, στην τροπολογία της Συμβαστική 9 έχουμε μια νέα διατύπωση για βέλτιστη ε, παροχή συμβουλών και προστασία ε, των δεδομένων. Στη Συμβαστική παρθμού 10 και έρχομαι τώρα στην ιδιωτική ζωή. Έχουμε μια νέα πρόταση για το πεδίο εφαρμογής, δύο προτάσεις για τη ασφάλεια που δέχτηκε, δηλαδή τις διαδικασίες ε, για την μη επιθυμητή ενημέρωση και πληροφόρηση. Όλα αυτά τα έχουμε συνεργαστεί με το Συμβούλιο και ε, θα ερχόμουν να προσθέσω και κάτι ακόμα εδώ. Στην πρώτη ανάγνωση ψηφίσαμε κάποια θέματα για την προστασία των δεδομένων και την παραβίαση και τα δέχτηκε όλα το Συμβούλιο, εκτό από ένα και αύριο θα ζητήσω να με υποστηρίξετε, να με το υπερψηφίσετε για να ενισχύσουμε τη θέση μα. Και τέλο, πρέπει να σα πω ότι κάναμε πολύ μεγάλη πρόοδο για τους καταναλωτές, ε, για την προστασία του στην ενιαία αγορά. Έχουν μπει τώρα ρυθμίσει στο κείμενο για την καλύτερη νομοθεσία την Πέμπτη το απόγευμα στις 4 η ώρα έχουμε νέο τριμερή διάλογο που σημαίνει ότι δεν θα είμαι σε όλη τη διακοινοβουλευτική διάσκεψη αλλά αυτό έχει προτεραιότητα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους και ηγητές μου και ελπίζω σε αυτή τη συνεδρίαση να κάνουμε σημαντική πρόοδο με το Συμβούλιο. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ήδη για τις ε, λεπτομέρειες. Στόχος μου είναι να ολοκληρώσουμε είτε αυτή την εβδομάδα, είτε πάρα πολύ σύντομα, εν πάση περιπτώσει, μετά τις ε, πασχαλινές διακοπές, για να έχω ένα συμβαστικό πακέτο πλήρες για την Ολομέλεια του Μαΐου, που θα είναι μεγάλη πρόοδος και επίτευγμα και πιστώνεται στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Συγγνώμη που μακρηγόρησα μάλλον, αλλά ήταν σημαντικό να εξηγήσω στους συναδέλφους ακριβώς περί τίνος πρόκειται και πού βρισκόμαστε σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Πολύ εμπεριστατωμένη η αναφορά σας. Δεν είναι κανένα από τους σκιώδεις εισηγητές εδώ. Θέλει άλλο συνάδελφος να κάνει σχόλια, δεν νομίζω. Σκιώδης ή μη σκιώδης. Η Κομισιόν θα ήθελε να μιλήσει ή το Συμβούλιο. Mr. Rodford, did you want to Η Προεδρία δεν είναι εδώ από το Συμβούλιο, αλλά η Κομισιόν είναι εδώ. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Χάρμπορ για αυτή την παρουσίαση της κατάστασης. Θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες με προσοχή. Ο κύριος Χάρμπορ ε, έχει δίκιο που είπε ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ σωστά εντόπισε τα κανθόδη θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στον τριμερή διάλογο. Θα προσπαθήσουμε να σα υποστηρίξουμε και στις λεπτομέρειες για να προχωρήσουμε. Γιατί το σημαντικό είναι να αποφύγουμε τη συνδιαλλαγή. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα στοιχεία για να αποφύγουμε τη συνδιαλλαγή. Κυρία Χάρμπορν, εσείς μιλήσατε με τους κοιόδες εισηγητές, όλοι τα ξέρουν λοιπόν όλα. Θα ψηφίσουμε αύριο ε, μία σειρά από συμβαστικές τροπολογίες. Θέλετε να κλείσουμε πριν περάσουμε στην παρουσίαση για το Solvit. Ο κατάλογος ψηφοφοριών ε, για την αυριανή ψηφοφορία είναι έτοιμος που δείχνει όλες τις, ε, τους συμβαστικούς ε, τομείς. Είναι οι τροπολογίες που θέλαν οι βουλευτές στη δεύτερη ανάγνωση αλλά όχι όλες. Δεν θα δεχτώ άλλες ε, τροπολογίες, γιατί αυτό που κάναμε τους κοινούς εισηγητές είναι να συμπεριλάβουμε όσο μπορούσαμε περισσότερο ε, τα θέματα στις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, επίσης, θα, με τις δικές μου τροπολογίες επαναφέρουμε και κάποιες βασικές τροπολογίες της πρώτης ανάγνωσης. Είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε μια βελτιωμένη πρόταση και είμαι χαρούμενος που το Συμβούλιο έδειξε διάθεση να διαπραγματευτεί και ευχαριστώ βεβαίως την Κομισιόν που μας βοήθησε στα δύσκολα θέματα. κυρίως για την ε, σύνταξη των τροπολογιών. Ε, σας, όπως είπατε, λέει Πρόεδρος, δεν θα δεχθούμε νέες τροπολογίες. Ελπίζω να είναι απλή η αυριανή ψηφοφορία και ελπίζω να είναι παρόντες και συνάδελφοι. Γιατί αλλιώς θα περάσουν η ψηφοφορία, ούτως ή άλλως, με εσάς ή χωρίς εσάς. Πάμε στο επόμενο σημείο που είναι ένα θέμα της κυρίας Ντέιλι, η οποία θα μας παρουσιάσει τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς και την έκθεση Solvit. Να σας υπενθυμίσω ότι η κυρία Σέντερσελτ έχει μια έκθεση δική της πρωτοβουλίας για τον πίνακα βαθμολογίας και ελπίζω η κυρία Ντέιλι να μας ενημερώσει για αυτές τις προτάσεις ούτως ώστε ε, η βουλευτής να τις λάβει υπόψη της, υπόψη της στις επόμενες εκδοχές του κειμένου. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε υπέρ του Solvit. Θέλουμε να λειτουργήσει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με το προσωπικό και την επάνδρωση των κέντρων Solvit. Ξέρω ότι οι πολίτες ε, εξακολουθούν να έχουν προβλήματα εφαρμογής νομοθεσίας. Ε, χαίρομαι λοιπόν για την υποστήριξη που τους δίνει και η υπηρεσία ανατολισμού των πολιτών ε, υπάρχει η ιδέα μιας ενιαίας πύλης, ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να παρουσιάζονται μέσα από μια και μόνη πύλη, φιλική για τους χρήστες, ε, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Παρακαλώ όσοι φεύγουν με ησυχία. Και αν θέλετε να μιλήσετε, έξω από την αίθουσα παρακαλώ. And as you can see, κυρία ότι μόνο οι καλοί μαθητές ε, έχουν παραμείνει στην αίθουσα. Εγώ θα πρέπει να χρειαστώ, ε, θα πρέπει να, φύγω για μια συνεδρίαση με τους ε, προέδρους των Επιτροπών. Ο κ. Μπουφών όμως θα προεδρεύσει τη θέση μου, θα του υποβάλλετε τα ερωτήματά σας και θα σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε, κυρία Ντέιλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μεγάλη μου τιμή που με προσκαλέσατε. Ποτέ δεν είχα έτσι το καινούριο κτίριο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Με μεγάλη χαρά το βλέπω για πρώτη φορά. Είναι σαφές για όλους μας πόσο σημαντική είναι η εσωτερική αγορά μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες και να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Όλα αυτά είναι σαφή. Αλλά με τη σημερινή κρίση είναι σαφές ότι θα πρέπει να τη φροντίσουμε την ε, εσωτερική αγορά. Αυτό που κάνουμε λοιπόν, ελπίζουμε, με τον πίνακα ε, βαθμολογίας της εσωτερικής αγοράς και με τον, την υπηρεσία προσανατολισμού των πολιτών και το Solvit είναι να τη βοηθήσουμε, να την πλαισιώσουμε την εσωτερική αγορά. Με βάση το τελευταίο πίνακα βαθμολογίας εσωτερικής αγοράς που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο, το μέσο κοινοτικό έλλειμμα μεταφοράς είναι 1% που είναι θυγραμμισμένο με το στόχο έλλειμματος μεταφοράς που καθορίζεται και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν διατηρήσει ή βελτιώσει τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν μια έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας εσωτερικής αγοράς. Παρ' όλα αυτά δεν το έχουν καταφέρει όλοι. Υπάρχει ένας μαυροπίνακας και ο μαυροπίνακας υπάρχει στη σελίδα 14 και 15 του πίνακα βαθμολογίας εσωτερικής αγοράς η εφαρμογή είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το θέμα δεν είναι να μεταφερθεί στην εσωτερική νομοθεσία έγκαιρα η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί και σωστά. Και εδώ έχουμε κάποια ανησυχητικά προβλήματα. Γιατί ο ρυθμός των ανοιχτών υποθέσεων επί παραβάση ε, παραμένει πεισματικά ψηλός. Ε, μπορούν Μπορεί να γίνει περαιτέρω οικονομική ενσωμάτωση, αλλά μόνο αν υπάρχει ισοτιμία στην αγορά. Στη σελίδα 16 μπορείτε να δείτε τις μεταβλητές που μας ανησυχούν σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας και μπορείτε να δείτε και το μαυροπίνακα που αφορά τις ανοιχτές υποθέσεις παραβάσεις σε σχέση με την ε, σωστή εφαρμογή του δικαίου. Δύο μαυροπίνακες λοιπόν τι οποίε μπορείτε να συμβουλευτείτε. Το άλλο πράγμα που κάναμε σε αυτόν τον πίνακα βαθμολογία είναι να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη μας κάποιες από τις συστάσεις της κυρίας Σέντεσορ και τη Έκθεση Ιδία πρωτοβουλίας της. Σε αυτό το πίνακα βαθμολογία λοιπόν εξετάσαμε τις εμπορικέ ροέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των τρίτων χωρών σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες και κεφάλαια βέβαια, τη ροή των κεφαλαίων. Για τα αγαθά, η αγορά είναι 16,9%. Ε, ενδοκινοτικά στις υπηρεσίες ε, το ποσοστό είναι 5% και σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές ροές στην Ένωση είναι 4%. Βλέπουμε από αυτά τα νούμερα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση στην εσωτερική μας αγορά. Και σε σχέση με τα αγαθά και σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα, και κεφάλαια βέβαια. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο πίνακα βαθμολογία εσωτερική αγορά να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την έγκαιρη μεταφορά τη κοινοτική νομοθεσία στην εσωτερική ένωμη τάξη και θα εξακολουθήσει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε λοιπόν είναι κάθε φορά που έχουμε ένα πίνακα βαθμολογία να λαμβάνουμε υπόψη και να εστιάζουμε σε διαφορετικού τομεί τη εσωτερική αγορά, Ελπίζω στον επόμενο πίνακα βαθμολογία, να ασχοληθούμε με τι δημόσιε προμήθειε και την εφαρμογή τη νομοθεσία στον τομέα αυτό σε όλε τις χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο θέμα αν λάβουμε υπόψη και το πακέτο οικονομικής τόνωσης που τα διάφορα κράτη-μέλη προωθούν. Ελπίζουμε λοιπόν στον επόμενο πίνακα βαθμολογίας ε, οι δημόσιες προμήθειες θα είναι το θέμα κλειδί. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε. Το άλλο είναι η ετήσια έκθεση του Solvit και το Κέντρο Προσανατολισμού των Πολιτών. Θα πω δύο λόγια για το καθένα. Θα ξεκινήσω με το Solvit. Το 2008 τα πήγαμε πάρα πολύ καλά σε επίπεδο Solvit οι υποθέσεις αυξήθηκαν κατά 22%, είναι τεράστια αύξηση και τώρα φτάσαμε το νούμερο ορόσημο χίλιες υποθέσεις το χρόνο. Οι περισσότερες προέρχονται από τους πολίτες. Το μερίδιο των επιχειρήσεων έχει μειωθεί κατά 14% στο 2008. Επομένως, υποθέσει από πολίτε αυξάνονται, υποθέσει από επιχειρήσει μειώνονται. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν εσεί ξέρετε γιατί. Αν έχετε κάποια στοιχεία που να δίνουν απαντήσει. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι τρέχει, τι υπάρχει πίσω από αυτή την αύξηση και τη μείωση. Και αν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια καλή στρατηγική για να καταπολεμήσουμε τη μείωση τη επιχειρήση. Στη Γενική Διεύθυνση Markt έχουμε αυτό το European Business Test Panel, όπου δίνουμε ερωτηματολόγια στις επιχειρήσεις ε, και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν μπορούν οι ίδιες επιχειρήσεις να μας δώσουν κάποιες ιδέες, γιατί δηλαδή, και να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί το solid δεν είναι πιο ελκυστικό στις επιχειρήσεις. Σε σχέση με τον αριθμό του 1000, ε, έχουμε πολύ καλό επίπεδο επίλυσης, 83%, αλλά έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Θα θυμάστε το προσωπικό προσλαμβάνεται από τα ίδια κράτη-μέλη και δουλεύει. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι των κρατών μελών αυτοί οι άνθρωποι. Κάθε κέντρο θα πρέπει να έχει 1,3 άτομα. Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Κάποια, πρέπει, δηλαδή, κάποια κέντρα θα πρέπει να έχουν ένα, ε, κάποια δύο και ο μέσος όρος είναι 1,3 άτομα. Αλλά τα μεγάλα κέντρα του Solvit, μιλάει για τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Αυστρία, δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πνιγμένοι μέσα σε βουνά υποθέσεων και δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το πρόβλημα. Νομίζω όμω ότι μπορούμε να πούμε ότι το Solvit χειρίστηκε περισσότερες υποθέσεις από τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές επί παραβάση. Επομένως, όντως κάνει κάτι το Solvit. Ε, είναι μια πολύ καλή εναλλακτική λύση για να ρυθμίσουμε το πρόβλημα της ε, λανθασμένης εφαρμογής του κοινωτικού δικαίου και να μειώσουμε τον όγκο των υποθέσεων του παραβάση. Επομένως, αυτό που λέμε στα κράτη-μέλη και αυτό που θα πείτε εσείς ελπίζω στα κράτη-μέλη είναι βοηθήσετε τα κέντρα Solvit, αυξήστε το προσωπικό τους, αυξήστε την ε, συνειδητοποίηση των επιχειρηματιών για τις ευκαιρίες και την ρεαλιστική προσέγγιση του Solvit. Το Solvit μπορεί να λύσει προβλήματα, υποθέσεις. Ένα άλλο πρόβλημα είναι, άλλο θέμα μάλλον, είναι ε, μια υπηρεσία ανατολισμού των πολιτών. Ε, είναι η υπηρεσία που την προσφέρει ένας εξωτερικός ανάδοχος που είναι ένα δίκτυο δικηγόρων σε όλα τα κράτη-μέλη που είναι εξειδικευμένοι στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται και στο ίντερνετ. από την Επιτροπή και διεκπαιρέωσε το 2008 11.000 υποθέσεις. Είναι φοβερό νούμερο. Πάνω από 90% από αυτές τις υποθέσεις διεκπαιρέωθηκαν μέσα σε τρεις μέρες. Απάντησαν δηλαδή οι δικηγόροι μέσα σε τρεις μέρες. Εγώ μίλησα ε, στους ανθρώπους στις δύο διαφορετικές αυτές υπηρεσίες ε, και μου είπαν ότι πραγματικά γνωρίζουν δυσκολίες οι πολίτες με την εσωτερική αγορά και ξέρουν πολύ καλά ποιες είναι οι δυσκολίες αυτές. Ε, οι τρεις προβληματικές περιοχές ήταν η κοινωνική ασφάλεια, τα επαγγελματικά προσόντα και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων το 2008 έτσι. Ήταν οι τρεις βασικοί τομείς, προβληματικοί τομείς θα έλεγα το 2008. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι αυτές οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, απαντούν στα προβλήματά τους. Και αυτό που ελπίζουμε είναι του χρόνου να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Να υπάρξουν περισσότερα ερωτήματα, περισσότερες υποθέσεις που θα επιλύσει το Κέντρο Προσανατολισμού των Πολιτών θα επιλύσει περισσότερες υποθέσεις το Solvit και θα υπάρξουν λιγότερες υποθέσεις όπου θα είμαστε αναγκασμένοι να σύρουμε τα κράτη-μέλη ε, στο δικαστήριο για λόγους παράβασης. Ευχαριστώ και θα απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσει. Ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίω και θα πρέπει να συγχαρούμε ότι συνάδελφο και κρίμα που είμαστε τόσο λίγοι εδώ μέσα. Το πρώτο που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επίτροπή Ευρωπαϊκής με οδηγεί στην εξή ερώτηση. Λέτε ότι ε, το δίκαιο μεταφέρεται με τρόπο ανεπαρκή. Ωραία. Και μη ικανοποιητικό. Αυτό το έχετε ε, ποσοτικοποιήσει, το έχετε μετρήσει. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν καλύτερα το δίκαιο. Και για το Σόλβιτ. τώρα έχω συγκεκριμένα μια ερώτηση. Μιλήσατε για χίλιες περιπτώσεις. Εγώ όταν απευθύνομαι στους Σλοβάκους πολίτες, δεν ξέρουν και πολλά πράγματα γι' αυτά. Στατιστικές έχετε εσείς. Οι περισσότερες περιπτώσεις του Σόρβιτ από ποια χώρα προέρχονται. Άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας μετέφερε όλες αυτές τις πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές για να έχουμε ακριβώς μία απογραφή ε, της κατάστασης. Ε, και ρωτώ, Κανονικά εμείς θα πρέπει να ε, αναγκάζουμε τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν καλύτερα ε, το κοινοτικό δίκαιο. Όχι μόνο να το μεταφέρουν ε, σωστά και καλύτερα, αλλά και το συντομότερο για να μπορούν οι πολίτες να υποφελούνται από όλα αυτά τα δικαιώματα που τους αναλογούν. Και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ερώτημα δεύτερο. Βεβαίω χρειάζεται αύξηση στους πόρους του Solvit, αυτό είναι προφανές. Αλλά εκεί δεν υπάρχει καμία αντένδειξη. Γιατί όσο καλύτερα δουλεύει το Solvit, τόσο περισσότερη ζήτηση έχει. Οπότε, μήπως είναι αντιφατικά αυτά που λέμε. Μια ερώτηση έτσι ανοιχτή, δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε, μπορεί να είναι ρητορική και αφορά εμένα προσωπικά. Μήπω το Solvit θα μπορούσε να είναι το κατεξοχή εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει ένας χώρος ουδέτερος. Δηλαδή, ζητούμε τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν έναν οργανισμό που έρχεται και τους αναγκάζει να εφαρμόζουν καλύτερα και να μεταφέρουν καλύτερα το δίκαιο. Μήπως να μας προβληματίσει αυτό. Uh, Μάλιστα. Δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Αν είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε και σε αυτό. Very interesting question. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Για την πρώτη ερώτηση. Αν έχουμε δηλαδή στη μελέτη που κάναμε στο πάνελ των επιχειρήσεων προγραμματίσει και αυτή την έννοια της μελέτης επιπτώσεων. Δηλαδή τι γίνεται όταν δεν μεταφέρουν την νομοθεσία, την κοινοτική τα κράτη-μέλη. Απάντηση όχι. Όχι σε αυτή τη μελέτη, αλλά το σκεφτόμαστε και μας απασχολεί. Διότι υπάρχει ένας τέτοιος κύκλος. Όταν κάποιος κάνει πρόταση νομοθεσίας και έχει και τον αντίκτυπο, στη συνέχεια, όταν φτάσουμε στο στάδιο που τα κράτη-μέλη δεν μεταφέρουν την νομοθεσία, τη μεταφέρουν εσφαλμένα, τότε υπάρχουν στοιχεία και δεδομένα ε, που να στοιχειοθετούν τη διαφορά μεταξύ των δύο. Αυτόν. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ε, εμείς κάνουμε προτάσεις συμβατές, αλλά τελικά ε, μετά τις διαπραγματεύσεις μπορεί να βγει τελείως διαφορετικό από εκείνο που προτείναμε εμείς διότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις ενημερώνουν εντός εισαγωγικών το πρόγραμμα αυτό, που δεν γίνεται πάντα. Για μας είναι λοιπόν διανοητική πρόκληση να προσπαθήσουμε να δούμε ποια ε, είναι η ε, μεταφορά και ποιος ο αντίκτυπος, αλλά προς τα εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούμε και να έχουμε σωστά στοιχεία γι' αυτό. Γιατί αυτό, έτσι πάει ο κύκλος ο λογικός. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. The statistics Οι στατιστικές για τη χρήση του Solvit είναι στην ίδια τη μελέτη, την έκθεση. Βλέπετε ότι κάποια κράτη-μέλη ανατρέχουν πολύ περισσότερο από μερικά. Αυτό έχει να κάνει αμυγός με τη διαφήμιση, την καλή, καλή τη συνειδητοποίηση του κοινού. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός δεδομένος που γενναιόδωρα μας έδωσε το Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητε αυτές και ζητήσαμε από τα διάφορα κράτη-μέλη και τις ομάδες του Solvit να κοιτάξουμε αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε για τη διαφημιστική εκστρατεία. Ορισμένοι είπαν ναι και διπλασίαστηκε ο φόρτος και άλλοι μας είπαν όχι προς Θεού γιατί έχουμε υπερβολικό φόρτο. Σε πρέπει λοιπόν κάθε φορά να βλέπουμε τι γίνεται επί στην εκάστοτε πραγματικότητα. Τώρα, σε έναν ιδανικό κόσμο, το θα είναι τόσο επιτυχές που θα καταργηθεί τελικά. Δηλαδή, σε ένα ιδανικό κόσμο θα έχουμε ένα στάδιο που δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα που να οφείλεται σε λάθος εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και εκεί θέλουμε να φτάσουμε, να αυτό καταργηθούμε. Ήμουν κάπου αλλού προηγουμένως στο Κοινοβούλιο και άκουσα ε, τι λένε τα κέντρα παροχή συμβουλών στους πολίτες παντού στην Ευρώπη και το ίδιο λένε και εκείνοι. Αν ε, συμβουλεύουμε αρκετά αρκετούς πολίτες και τελικά αυτά μεταφέρονται στις κυβερνήσεις, να δούμε τι πάει στραβά, τότε κάποια στιγμή δεν θα χρειαστούμε πια και θα καταργηθούμε. Αυτό είναι η ύψιστη αξιολόγηση δηλαδή της ε, επιτυχίας. Σωμάς τεχνικ, έτσι το λένε, δηλαδή να είμαστε σε διαθεσιμότητα τελικά ακριβώς επειδή δεν μας χρειάζεται. Βέβαια έχει πόρο αυτή η κατάσταση. Και αν δούμε τι γίνεται με την νομοθεσία που προετοιμάζεται τώρα στην εσωτερική αγορά και πρέπει να μεταφερθεί στα κράτη-μέλη μέχρι το 2010, εκεί να δείτε χιονοστιβάδα, τσουνάμι προβλημάτων αναμένεται στα κέντρα Solvit. Ρωτήσατε επίσης αν θέλουμε το Solvit να είναι ένα εργαλείο πανευρωπαϊκό και όχι των κρατών μέλων. Η απάντηση είναι όχι, σε καμία περίπτωση, διότι Αυτό που είναι το ωραίο στο Solvit είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλάβουν ότι εφαρμόζουν λάθος την κοινοτική νομοθεσία. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη και ο, ο κόσμος επιτόπου, ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπηρεσίες να συνεργάζονται για να εφαρμόζονται σωστά τα προγράμματα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι ο μαύρος κακός λύκος αυτή την ιστορία. και έχει ναρόπολα και χτυπάει τα κράτη-μέλη. Η διαδικασία προσφυγής επί παραλήψη χρειάζεται δύο χρόνια και μέχρι να ε, παραπευθούν τα κράτη στα δικαστήρια και να τελεσιδικήσει υπόθεση μπορεί να περάσουν και πέντε χρόνια. Εμείς για να λύσουμε ένα πρόβλημα χρειαζόμαστε πέντε χρόνια, ενώ τα κράτη-μέλη μπορούν να το λύσουν μέσα σε δέκα εβδομάδες. Οπότε το Solvit δεν μπορεί να είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μέγα ευεργέτημα από το Solvit είναι ότι συνεργάζονται οι διοικήσεις, τα κράτη-μέλη. Και εκεί θα πρέπει να δούμε και τους πολίτες και το Solvit να έχουν κοινό σεμινάριο για να συνεργάζονται. Έχετε προσκληθεί κιόλα σε ένα πρόγευμα εργασία και χαίρομαι που θα έρθετε να τους συναντήσετε. Α, κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον εδώ. έχουν συνεργαστεί ως ε, δίκτυο έτσι, για να λύνουν τα προβλήματα. Είναι θαυμάσιο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει δίκτυο εθνικό και κέντρο για την επίλυση προβλημάτων. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Χάρμπορ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε. Αλλά έπρεπε να λύσω κάποια προβλήματα για την αυριανή ψηφοφορία, οπότε δεν άκουσα αυτά τα οποία είπατε, αλλά έχω διαβάσει τα έγγραφα. Ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα για τα κέντρα πληροφόρησης και ειδικά για το σύστημα πληροφόρησης εσωτερικής αγοράς. Γιατί νομίζω πως είχατε δίκιο πριν όταν είπατε πόσο κρίσιμη είναι η παροχή πληροφοριών στους πολίτες επιχειρήσεις αλλά καθώς προχωράμε και με την οδηγία των υπηρεσιών έχουμε και μια διαδικασία ελέγχου, δηλαδή οι διοικήσει ανταλλάσσουν στοιχεία που θα οδηγήσει σε πιο συνεκτική εφαρμογή της οδηγίας. Είχαμε και μια συζήτηση με τον κύριο Φερχόγγεν πριν. Οι διατάξεις του πακέτου για τα εμπορεύματα επίσης ε, συνδέονται και με τις ε, πληροφορίες και δεδομένου του ότι αφορά αυτό και υπηρεσίες και παραγωγή δηλαδή Ένας παραγωγός θα πρέπει να στείλει επαγγελματίε σε άλλη χώρα να εγκαταστήσουν το σύστημα κτλ δεδομένων όλων αυτών θεωρείτε ότι ίσως ε, στον επόμενο, με την επόμενη κομισιόν θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σε κάθε πτυχή της εσωτερικής αγοράς για να προχωρήσει αυτό το θέμα. Γιατί αυτή μου φαίνεται ότι είναι η επόμενη λογική εξέλιξη για να γίνει η πολιτική της ε, ενιαίας αγοράς ολοκληρωμένη. Επίση, δεν ξέρω γιατί είναι το σύστημα εσωτερικής πληροφόρησης εσωτερικής αγοράς και όχι ενιαίας αγοράς, αλλά εν πάση περιπτώσει. You always ask me such hard questions. δύσκολες οι ερωτήσεις, δύσκολες. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, Η αμοιβή αξιολόγηση της οδηγία των υπηρεσιών από τα κράτη-μέλη θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί εκεί θα δούμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο το ποιε απαιτήσει είναι εύκολο να εκπληρωθούν και ποιε όχι. Και επειδή αυτό γίνεται ταυτόχρονα ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί και η οδηγία και να αρχίσουν να κινούνται οι υπηρεσίε Οπότε ταυτόχρονα είπα πως θα έχουμε ένα τσουνάμι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπερέβαλα, θα έχουμε δύο κύματα ετοιμάτων. Θα έχουμε ένα κύμα ετοιμάτων που θα είναι εσωτερικό στην δημόσια διοίκηση, όπου θα ρωτάνε μεταξύ τους και η Κομισιόν θα ζητάει πληροφορίες. Ε, αυτό θα πρέπει να περάσει μέσα από το, ε, το ηλεκτρονικό αυτό λογισμικό το ένα επίπεδο είναι αυτό και σε ένα άλλο επίπεδο οι ίδιες οι υπηρεσίες και τα άτομα που θέλουν να απασχοληθούν σε αυτό το τομέα να περνάνε από το Solvit ε, και τις υπηρεσίες των πολιτών ε, και τη διεύθυνση επιχειρήσεων και το Your Europe, όλοι αυτοί θα έχουν τα ίδια Οπότε, Ε, ελπίζουμε ότι θα έρθει έτσι ώστε η επιφύρηση η λογική του να έχουμε μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Οπότε προσπαθήσαμε τουλάχιστον οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της ενιαίας αγοράς να συνεργαστούν ε, με υπ' αυτή την ε, ορολογία που λέμε SMAS, δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες της ενιαίας αγοράς έτσι ώστε ανεξαρτήτως ε, του πού θα απευθυνθεί στην Κομισιόν ένα άτομο ή μια επιχείρηση θα λάβει την ίδια απάντηση. Και εμείς θα λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο. Και είχαμε, είχα κάνει εγώ μια ωραιότατη παρουσίαση με ένα στόχο για βελάκια. Για να δείξω ότι πρέπει όλοι να έχουμε έτσι, τον ίδιο στόχο. 2010. Για να επιτύχουμε έτσι. Το εξή στόχο, ανεξαρτήτως του πού θα απευθυνθεί κανείς, να είναι ίδιο το αποτέλεσμα στην πλευρά της, ε, της ζήτησης. Και αν τα καταφέρουμε από αυτή την πλευρά, οπωσδήποτε και τα κράτη-μέλη από την περιά της ε, παροχής θα μπορούν να το κάνουν. Αλλά αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα. Είναι σοβαρό είναι μια πρόκληση. Και άλλο θέλει το λόγο. Όχι. Χαίρομαι που συγκράτησα δύο πράγματα ε, ε, σήμερα. Το ένα είναι ε, δίκτυα εταιρική σχέσης που γεννιούνται και αυξάνονται και χαίρομαι. Και το δεύτερο, ο στόχος αυτός ότι ο στόχος μιας διοίκησης είναι να πετύχει και τελικά να αυτοκαταργηθεί. Αυτό είναι για μένα συναρπαστική ιδέα. Και ε, σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε. Κυρίσω το πέρας της συνεδρίασης. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.